Pour euh, ce retard, mais euh, Θα ασχοληθούμε, θα ακολουθήσουμε την ε, ημερήσια διάταξη. Έχουμε μία μικρή καθυστέρηση. Θα ασχοληθούμε με το θέμα του αυταρχισμού και την περιστολή ελευθερίας και έκφρασης με τρεις ε, περιπτώσεις και μελέτες για την Κίνα, Αίγυπτο και Ρωσία. Δεν ε, έχουμε επιλέξει αυτές τις χώρες ε, τυχαία, αλλά εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει καταστολή της ελευθερίας τύπου και των ελευθεριών. Γι' αυτό στους συντονιστές αποφασίσαμε να στοχεύσουμε στις τρεις αυτές χώρες που γνωρίζουν μία ιδιάζουσα κατάσταση και έχουμε καλέσει πρόσωπα που θα μας ε, ε, διευκρινίσουν την κατάσταση. Δεν θα μακρηγορήσω, θα δώσω το λόγο στον Κλεμά, Κλεμά Νιαλέτσόση Βουλέ, εάν ε, έχω προφέρει σωστά το όνομά σας που ασχολείστε, είσαστε ειδικό εισηγητής από τα Ηνωμένα Έθνη για το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε και συνέρχεστε. Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που με καλέσατε να αναφερθώ στο ζήτημα αυτό έχω υπάρξει ειδικό εισηγητής ε, του ΟΗΕ για το δικαίωμα του συνέργεστε από το 2018. Έχουμε εντολή να αναφέρουμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για αυτά τα δικαιώματα ανά τον κόσμο. Ως εισηγητής ε, καθήκον μου είναι να εξετάζω προσεκτικά το περιβάλλον εντός του οποίου λειτουργεί η κοινωνία των πολιτών ε, και βλέπω ότι γίνεται όλο και πιο περιοριστικό. Καλώς όρισε την ευκαιρία αυτή που έχω να μοιραστώ μαζί σας ε, το πώς ε, το ζουν αυτό οι άνθρωποι επιτόπου. Κυρίε και κύριοι βουλευτές, τα δικαιώματα του συνέρχεστε ειρηνικά είναι βασικό μέρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βασικό συντελεστής της ανάπτυξης και της δημοκρατίας. και έτσι ο κόσμος ε, μπορεί να επιδιώκει κοινού ε, σκοπούς ε, και δίνει την ευκαιρία να εκφραστούν οι αντιφρονούντες, να μετασχηματίσουν τον κόσμο, να επισημάνουν διάφορες καταστάσεις και να διαμορφώσουν το μέλλον. Από όταν ορίστηκα έχω δει την δύναμη που μπορεί να έχει η κοινωνία των πολιτών στην ε, ειρηνική πρόοδο της ε, κοινωνίας. Μπορώ να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Αρμενία, την Ισία, όπου χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα δικαιώματα την κοινωνία των πολιτών για να προωθήσουν την αλλαγή. Μπορούμε να σας δώσουμε και τα παραδείγματα του Σουδάν, όπου είχαμε κάποιους ε, θανάτους. Και μπορούμε επίσης να δώσουμε και το παράδειγμα του κινήματος ΜΗΤΟΥ ε, αλλά και την κλιματική απεργία των παιδιών ανά τον κόσμο. Δυστυχώς όμως ε, τα δικαιώματα αυτά του συνέρχεστε υφίστανται μία επίθεση. Βλέπουμε μία οπισθοχώρηση των δικαιωμάτων αυτών. Ε, καταστολή, ποινικοποίηση, και εκφοβισμό κατά των ηγετών της κοινωνίας των πολιτών. Βλέπουμε το πώς οι παλαιές και νέες τακτικές καταστολής χρησιμοποιούνται ε, βία κατά των διαδηλωτών, κλείσιμο του διαδικτύου για να ενσπείρουν τον φόβο. Επίσης βλέπουμε το πώς ε, αυξάνεται ο απολυταρχισμός και υπάρχει μια ρητορική κατά των δικαιωμάτων ανά τον ε, κόσμο. Και έχουμε επιθέσεις κατά των ατόμων που υπερασπίζουν τα δικαιώματα αυτά. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, στην ε, πρώτη μου έκθεση προς το 38, 38 ε, Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξέτασα ποιες ήταν οι μεγαλύτερες παγκόσμιες τάσεις που εμπόδιζαν την εξάσκηση των δικαιωμάτων αυτών. Στην ακρόαση αυτή θα ήθελα να επισημάνω τρεις ε, μεγάλες ε, τάσεις που θεωρώ ότι έχουν σημασία για το σημερινό μας θέμα. Πρώτα είναι η χρήση της νομοθεσίας για την καταστολή του δικαιώματος του συνέρχεστε. Η καταστολή δηλαδή η υπομορφή νομοθεσίας είναι το εργαλείο της νέας απολυταρχίας με μια επίφαση νομιμότητας πάρα πολλές κυβερνήσεις ανά τον κόσμο απειλούν την ύπαρξη της κοινωνίας των πολιτών. Νόμοι οι οποίοι εμποδίζουν το σχηματισμό και την καταγραφή και τη λειτουργία των διαφόρων ενώσεων, όπως αυτός ο οποίος εγκρίθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στη Γουατεμάλα, που επιβάλλει ε, βαρύτατους περιορισμούς ε, στην χρηματοδότηση, ειδικά από το εξωτερικό. Νόμους που απειλούν ε, τους ηγέτες κοινωνίας των πολιτών ποινικέ διώξεις που καθιστούν ε, τους οργανώσεις αυτές ε, αντικείμενα αυθαίρετων διώξεων. Επίσης βλέπουμε πως αυξάνονται τα εμπόδια. Υπάρχουν γενικές απαγορεύσεις, γεωγραφικοί περιορισμοί, υποχρεωτική αδειοδότηση, ε, νομικά μέτρα δηλαδή. Δεύτερον, υπάρχει η ποινικοποίηση της ειρηνικής διαμαρτυρίας και η αδιάκριτη χρήση βίας για την καταστολή που αποτελεί ένα άλλο ε, σημάδι και σε δημοκρατικές και σε αυταρχικές ε, χώρες, οπωσδήποτε περισσότερο στις δεύτερες. Συνελεύσεις και διαμαρτυρίες ε, θεωρούνται απειλή κατά της εθνικής ασφαλείας. Οι εθνικές αρχές ανταποκρίνονται με βία και με το βαρύ χέρι του ποινικού δικαίου. Συγκεκριμένα τη αντρομοκρατικής νομοθεσίας έχουμε δει επίση κράτηση και βασανιστήρια διαδηλωτών. Πολλών με ψευδείς κατηγορίες. Τα δε κράτη τα τελευταία χρόνια δεν εμφανίζονται τόσο διατεθειμένα να εμπλακούν σε διάλογο. Τρίτον, υπάρχουν οι περιορισμοί στην άσκηση των ελευθεριών αυτών, του συνέρχεστε και του συνεταιρίζεστε και στο διαδίκτυο. Παρατηρούμε διάφορες απαγορεύσεις ε, πρόσβασης σε διάφορες πλατφόρμες, σε κοινωνικά μέσα αυστηρές ποινές για τη δημοσίευση των λεγόμενων ψευδών ειδήσεων ή δυσυμιστικού περιεχομένου και ευρύτατες διατάξεις ε, που υπάρχουν σε νόμους περί κυβερνοεγκλήματος. Βλέπουμε πολύ προχωρημένα εργαλεία ψηφιακής παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται κατά της κοινωνίας των πολιτών χωρίς καμία λογοδοσία. Βλέπουμε πως τα εργαλεία αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε δολοφονία των ανθρώπων αυτών το συχνό κλείσιμο του διαδικτύου και εκστρατείες παραπληροφόρησης χρησιμοποιούνται για να καταστήλουν τις ε, κοινότητες και να διασπείρουν σύγχυση. Κυρίε και κύριοι βουλευτές, τα τελευταία χρόνια έχουμε δει σοβαρές προσπάθειες από την διεθνή κοινότητα για να αντιστραφούν αυτές οι τάσεις. Παραδείγματο χάρη η εντολή που μου ανατέθηκε πριν από 10 χρόνια Έχουμε κάνει επισκέψεις σε 13 ε, χώρες ε, και έχουμε κάνει τις ανάλογες συστάσεις. Έχουμε στείλει πάνω από χίλιες ανακοινώσεις για διάφορες χώρες. Έχουμε εκδώσει 16 θεματικές εκθέσεις και έχουμε κάνει σημαντικές διαβουλεύσεις ανά τον κόσμο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Ένωση για την στήριξη που έδωσαν στην εντολή αυτή τα χρόνια αυτά. Αλλά ε, βρισκόμαστε το μέσο ενός παγκόσμιου αγώνα για το μέλλον της ισότητας του πλανήτη και των δημοκρατικών αξιών μας. Σε τέτοιους καιρούς ακριβώ χρειάζονται τα δικαιώματα του συνέρχεστε έτσι ώστε ο κόσμος να μπορεί να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του και να διαμορφώσει το μέλλον του. Κυρίε και κύριοι βουλευτές, τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι σημαντικό να στηρίξουμε την κοινωνία των πολιτών κατά των πιέσεων αυτών. Όλες οι προσπάθειες αυτές που γίνονται για να αποθηθεί η ε, περιοριστική νομοθεσία πρέπει να ενισχυθούν. Η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για να εφαρμοστούν σωστά οι διεθνείς κανόνες. Εξάλλου, αυτοί μπορούν να αλλάξουν την τοπική πραγματικότητα. Επίσης, να γεφυρώσουμε το κοινό μεταξύ κοινωνικών κινημάτων και παραδοσιακών υπερασπιστών ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να γεφυρώσουμε το κενό αυτό, έτσι ώστε να προστατεύονται τα μέλη των κοινωνικών κινημάτων, να έχουν νομική και άλλη αρρωγή, αν υπάρχει καταστολή, και να μπορούν ε, να αναπτύσσουν τα επιχειρήματά τους με όρους ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις υποχρεώσεις των κρατών. των κρατών. Σημαντικό είναι επίσης να προστατεύσουμε το διεθνέ σύστημα, ειδικά το σύστημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατά των επιθέσεων που βλέπουμε και τη ρητορική που προσπαθεί να τους απονομιμοποιήσει. Θα πρέπει επίσης ε, να σχετίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα με την ανάπτυξη και θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνουμε το διάλογο μεταξύ όλων των μερών μεταξύ ε, διαφόρων πλευρών για να βρεθούν αποτελεσματικές λύσεις σε τοπικά και παγκόσμια προβλήματα. Πρόκειται για μια ατζέντα για ένα πρόγραμμα πολύ φιλόδοξο, το οποίο είμαι προσελωμένος, αλλά για να πετύχει βεβαίως χρειαζόμαστε και τις δημοκρατικές κυβερνήσεις. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει ηγετικό ρόλο στα θέματα αυτά. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ηγηθεί ως ομάδα στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά το πιο σημαντικό πρέπει να συνεχίσει να βοηθά τα μέλη της κοινωνίας των πολιτών, τον κόσμο. Ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να σας δώσω απευθεία το λόγο γιατί ξέρω ότι πρέπει να φύγετε νωρίτερα. Εάν τα μέλη λοιπόν έχουν ερωτήσεις, για την πρώτη παρουσίαση. Παρακαλώ, Ιζαμπέλ. Καταρχήν θα ήθελα να χαιρετήσω τον καλεσμένο μας και να πω ότι συμμερίζομαι τις σκέψεις του για τη σημασία της κοινωνίας των πολιτών μέσα στα πλαίσια ενός κοινωνικού και ευρωπαϊκού που γίγνεστε για την προστασία των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατανοώ τις ανησυχίες του για τον εγκληματικό χαρακτήρα που δίνουν οι κυβερνήσεις στην κοινωνία των πολιτών καθώς και τους κοινωνικούς κλειδονισμούς στις διάφορες χώρες οι οποίοι καταστέλλονται και να τονίσω την ύπαρξη του νόμου κατά της ε, τρομοκρατίας που χρησιμοποιείται καταχρηστικά για να πλήξει τους ακτιβιστές σε όλα τα σημεία του κόσμου όπου χρησιμοποιείται ο εκφοβισμός και η τρομοκρατία για να προωθηθεί η καταστολή. Οι δημοκρατικές κοινωνίες γνωρίζουν μια μεγάλη κρίση, ενώ τα πολιταρχικά καθεστώτα ε, δυστυχώς αναδύονται. Αυτό συμβαίνει και γι' αυτό θα πρέπει να μην θεωρήσουμε κάτι δεδομένο τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι κάτι που θα πρέπει να απασχολεί καθημερινά και να δίνουμε μεγάλες μάχες. Άκουσα για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς θεωρείτε εσείς ότι πρέπει να γίνει μια εντατικοποίηση δραστηριότητας. Πώς θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να κατέχει ηγετικό ρόλο στον κόσμο για την πρόσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να σας υποβάλω μία ερώτηση όταν μιλήσατε για το ρόλο της Ευρώπης που είναι η κινητήρια δύναμη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ε, κατά της καταστολής. Υπάρχουν πολλοί παρατηρητές που ασχολούνται με τον πολύπλευρο χαρακτήρα του εμπορίου. Πολλοί βεβαίως θεωρούν ότι δεν υπάρχει αυτός ο πολύπλευρος χαρακτήρας στη, στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά μας λένε τα Ηνωμένα Έθνη. Θεωρείται λοιπόν ότι ορισμένες χώρες τα Ηνωμένα Έθνη δεν προασπίζονται αυτά τα δικαιώματα. Και πώς βλέπετε το ρόλο της Ευρώπης στα Ηνωμένα Έθνη έναντι χωρών που έχουν μία προσέγγιση πολιτισμικού σχετικισμού. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις δύο αυτές ερωτήσεις που πάνε στην καρδιά μίας από τις πτυχές που έφυξα στην παρουσίασή μου. Καταρχά είναι σημαντικό σήμερα έναντι όλης αυτής της αμφισβήτησης των αρχών, των αξιών της δημοκρατίας και της καταπίεσης που υπάρχει. Οι χώρες που έχουν βασίσει την παράδοσή τους, το σύστημά τους οι χώρες που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτήν την άνοδο της απολυταρχίας της καταπίεσης. Σήμερα που ασκούνται επικρίσεις το διεθνές σύστημα που το διεθνές σύστημα υφίσταται επιθέσεις μάλιστα αλλά που όλοι εμείς εδώ γνωρίζουμε ότι αυτό το σύστημα το φτιάξαμε μετά από μεγάλες θυσίες. Ε, συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει αυτό το σύστημα να καταστεί πιο αποτελεσματικό, αλλά οι χώρες που προσπαθούν να καταστρέψουν το σύστημα έχουν πολύ συγκεκριμένες και κρυφές, τα έλεγα, στοχεύσεις. Σήμερα ως ειδικό συγητής έχω τις δικές μου συστάσεις, έχω τις δικές μου ιδέες για το τι πρέπει να κάνουμε για να βελτιώσουμε, να ενισχύσουμε το σύστημα και εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να βελτιώσουμε μια σειρά από πράγματα, αλλά δεν μπορούμε απλά σήμερα να πετάξουμε αυτό το σύστημα στον κάλαθο των αχρήστων. Γιατί μας επέτρεψε να κάνουμε κάποια βήματα προς τα εμπρός. Μιλούμε για ένα σύστημα προς το οποίο στο οποίο έχουν προσχωρήσει ένα μεγάλος αριθμός χωρών στον κόσμο. Δεν πρέπει να αφήσουμε λοιπόν να εξαφανιστεί ή να καταστραφεί και θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι ηγέτιδα στην προσπάθεια αυτή υπεράσπισης ότι δηλαδή η ελευθερία έκφρασης, η ελευθερία του συνεταιρίζεστε, του συνέρχεστε πρέπει να είναι βασικές αρχές Τη υπεράσπισης αυτής, τη άμυνας αυτή του συστήματος. Είναι λυπηρό ότι όλο και πιο συχνά είναι δυσδιάκριτη η φωνή η τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ενιαία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί επαναλαμβάνω σήμερα πλήττεται η δημοκρατία η πιο σημαντικές ανθρώπινες αξίες. Επομένως πρέπει η κάθε χώρα να αφήσει τα μέρος της, ε, τα συμφέροντα, τα τοπικά δικά της συμφέροντα, για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την εκστρατεία καταπίεσης, καταστολής που στοχεύει στην καταστροφή του δημοκρατικού συστήματος και του κοινού χώρου που έχουμε να συζητούμε. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Θα περάσουμε τώρα στο, στο σημείο το πιο συγκεκριμένο αναχώρα. Έχουμε τον κύριο Γιάν Λι Γιάνγκ, που είναι επικεφαλής του China Citizens Power, ηγέτης ε, του κινήματος εκδημοκράτησης της Κίνας, ε, πρώην κρατούμενος του καθεστώτος ε, από το 2002 στο 2007 σύμπροεδρος της διακήρυξης της Γενέβης για την ελευθερία του διαδικτύου το 2010 έλαβε διάφορες διεθνείς βραβεύσεις Harvard Alumni Achievement Award μεταξύ άλλων έχετε το λόγο ε, δεν ξέρω αν με ακούτε κύριε Young έχετε το λόγο για 10 περίπου λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε σε αυτήν την απολύτως επίκαιρη και σημαντική συνεδρίαση. Επίκαιρη διότι η πανδημία του κορονοϊού έχει καταδείξει τις ε, πολύ επικίνδυνες ελλείψεις ε, του απολυταρχικού καθεστώτος ε, της λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας υπό τον Σι ε, Jinping. Η κακή διαχείριση, η ελλειπής διαχείριση της κατάστασης, της κρίσης από το καθεστώς και οι επιπτώσεις για το σύνολο της κινέζικης κοινωνίας σχετίζονται απολύτως με τις απολυταρχικές πολιτικές που ακολουθεί ο ίδιος ο ΣΥ. όλα αυτά που θα μπορούσαν να πάνε άσχημα υπό την κρίση αυτή, υπό την έκρηξη αυτή, πήγαν άσχημα υπό την ηγεσία του Xi Και είναι ακόμα χειρότερα υπό τη δική του ηγεσία, διότι έχει αναλάβει όλο τον έλεγχο του κόμματος και του κράτους, συμπεριλαμβανομένης της ηγεσία του στρατού, των ενόπλων δυνάμεων και της αστυνομίας. Έχει την απόλυτη εξουσία στην οικονομική πολιτική, που είχε ανατεθεί στο κόμμα από τη δεκαετία του 80 και εντός του κόμματος ο ΣΥ λειτουργεί σαν να είναι αφεντικό σε όλα. Ο έλεγχος του των ενόπλων δυνάμεων είναι ακόμα πιο πλήρης και απόλυτος από ότι εκείνος που ασκεί στο κόμμα και στην κυβέρνηση. προσπαθεί να εξασφαλίσει απόλυτη αφοσίωση στο κόμμα και στον εαυτόν του και τα μέλη του κόμματος ε, έχουν αυστηρές οδηγίες να αποφεύγουν οποιαδήποτε ακατάλληλη συζήτηση, οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή αμφιβολία. Διατηρεί το κόμμα στην γραμμή που έχει επιλέξει ο ίδιος και υποσκάπτει και αφαιρεί τη δυνατότητα οποιοδήποτε άλλου πολιτικού, οποιοδήποτε άλλου πολίτη να αμφισβητήσει την απόλυτη εξουσία του. Επίσης έχει κάνει μια ιδεολογική στροφή προς τα αριστερά, λέει ο Μίλτης, σκορπώντας τον δρόμο σε ακαδημαϊκούς, δημοσιογράφους και επιχειρηματίες. Έχει επιστρέψει σε μια τρομοκρατία τύπου ΜΑΟ, και θέλει να ελέγχει όλα τα στοιχεία της ζωής των πολιτών στην Κίνα. Στο 19ο συνέδριο του κόμματος, που ξεκίνησε και η δεύτερη θητεία του ΣΥ, ξεκίνησε αναφέροντας ένα διάσημο ρητό του ΜΑΟ. Κόμμα, κυβέρνηση, στρατός, ακαδημία, πολίτες, Ανατολή, Δύση, Βορράς, Νότος, Κέντρο, το κόμμα, ηγείται των πάντων. Πέραν της απόλυτης πολιτικής ε, εξουσίας, εξασφαλίζεται ότι το, το κόμμα έχει το απόλυτο μονοπόλιο στον οικονομικό τομέα. Υπό τον ΣΥ, η διατήρηση της σταθερότητας και ο κρατικός μηχανισμός έχει γίνει ακόμη πιο αποτελεσματικός και απολυταρχικός. Δεν υπάρχουν πλέον το παραμικρό κενό, το παραμικρό ρήγμα διαρροής πληροφοριών που θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί οποιοδήποτε που θα ήθελε να ενημερώσει την κοινή γνώμη. Όλα είναι κεντρικοποιημένα και ο ΣΥ ε, λέγει, δηλώνει πως βρίσκεται σε έναν αγώνα για τον έλεγχο της κοινή γνώμης. Πάνω από 30.000 ε, κινέζικες επιχειρήσεις παρακολούθησης έχουν πάνω από 1,5 εκατομμύριο υπαλλήλους. Μεταξύ άλλων η Huawei, η, η Dahua και η Hikvision. Τα προϊόντα όπως το Hikvision, ή μάλλον οι κάμερες της Hikvision, πολλούνται ευρύτατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποιες επιχειρήσεις όπως η Alibaba και η Tencent ε, χρησιμοποιούν την ελεύθερη αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να έχουν πρόσβαση στο κεφάλαιο και στην τεχνολογία ώστε να αναπτύξουν περισσότερα προϊόντα παρακολούθησης. Όλο αυτό το σύστημα παρακολούθησης επιτρέπει στην Κίνα να έχει οικονομήσει ένα τεράστιο δίκτυο παρακολούθησης και όπως και στην ωκεανία του Όργουελ η βαθύτερη αιτία είναι να προλάβουν οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή κίνδυνο για την απόλυτη εξουσία του κόμματος. προκειμένου να βελτιώσουν, όπως λένε οι ίδιοι, την τρισδιάστατη νομιμοποίηση, εξειδίκευση και ευφυΐα της ε, κοινωνικής πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλειας. Και τώρα η το σύστημα αυτό παρακολούθηση, εκτείνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Ο μεγάλος στόχος της ε, ανανέωσης το όραμα του κινέζικου κράτους επιτρέπει το κράτος κόμμα αυτό να συνεχίσει να αρνείται τα πολιτικά δικαιώματα των Κινέζων υπηκόων όπως και των κατοίκων του Χονγκ Κόνγκ λέει ο μιλτής, να ελέγχουν απολύτως ε, τους πληθυσμού στο Θιβέτ και τους μουσουλμανικούς πληθυσμού στο Ουιγκούρ και παραβιάζουν κάθε αρχή χρηστής διακυβέρνησης με βία και με τρομοκρατία. Ο υπόλοιπος κόσμος κοιτάζει προς την Κίνα και περιμένει μια εναλλακτική, ένα ενελικτικό πρότυπο διακυβέρνησης, αλλά κινείται ο κόσμος προς το, προς το μοντέλο του ένας κόσμος δύο συστήματα. Με απευθείας ανταγωνισμό προς την φιλελεύθερη δημοκρατία πλέον παραδέχεται ανοιχτά η Κίνα την αναπόφευκτη άνοδο και επικυριαρχία της ονειρεύεται είναι ότι θα οδηγήσει τον υπόλοιπο κόσμο προς το μέλλον. Και η μεγάλη αυτή στρατηγική προσπαθεί να αποφύγει την άμεση αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να εκμεταλλευτεί τις, την ύπεθρο του κόσμου, την επαρχία του κόσμου, τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, ώστε να αναπτύξει μια στρατηγική κατά των ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βασικό πεδίο μάχης για την παγκόσμια κυριαρχία που, επιχειρεί η Κίνα. Η πρόκληση είναι τα ψέματα, οι ψευδείς θέσεις και τοποθετήσεις της ε, κυβέρνησης της Κίνας και η προσποιούμενη υιοθέτηση κάποιων από τις δυτικές ε, φιλελεύθερες αρχές προκειμένου να κερδίσει τον τελικό αγώνα. Παρουσιάζονται ως ειρηνικοί απολυταρχικοί ηγέτες για να επεκτείνουν την επιρροή τους στην Ευρώπη. Η κεντρική Ευρώπη είναι ιδιαίτερο στόχος διότι η Κίνα πιστεύει ότι αυτή η περιοχή είναι ασθενής κρίκος όπου η δημοκρατία δεν είναι απολύτως ριζωμένη. Πιστεύουν ότι εκεί μπορούν να πετύχουν πολλά. Επίσης προσπαθούν να επιτύχουν την επικυριαρχία του κινέζικου νομίσματος έναντι του δολαρίου, λέει ο μιλτής. Άλλη μια στρατηγική είναι η χρησιμοποίηση της τεχνολογίας του 5G από τη Huawei. Αυτά που σημαίνουν όλα αυτά για τον κόσμο είναι ότι η Κίνα βρίσκεται σε επιθετική στάση, επιτίθεται αυτή τη στιγμή με την πρωτοβουλία Road and Belt, έργα υποδομών μεγάλης κλίμακας, την Τράπεζα Επενδύσεων και Υποδομών, το όραμα της Κίνας για, την, για, την, για το κοινό πεπρωμένο της ανθρωπότητας. Παρά τις φιλοδοξίες ε, παγκοσμίου εμβελίας της Κίνας και την επιθετική της εκστρατεία, η αποτυχία του καθεστώτος στον έλεγχο της πανδημίας του Βουχάν είναι προφανής. Ο ιός έχει ταράξει τον έλεγχο, την εξουσία του Xi Jinping. Στις 6 Δεκεμβρίου του 2012, πριν από 7 χρόνια, κύριε Πρόεδρε, είχα μιλήσει σε μία ακρόαση στην ίδια δική σας υποεπτροπή και είχα προβλέψει τότε ότι δεν θα υπάρξει κάποια ουσιαστική αλλαγή στο απολυταρχικό καθεστώτος Κίνας στα επόμενα τρία χρόνια, αλλά μάλλον θα υπάρξει μια σημαντική αλλαγή τα επόμενα 5 με 10 χρόνια. Ίσως τότε να είχα εκπλήξει αρκετούς συναδέλφους σας λέγοντας αυτό, αλλά είχα βασιστεί στην ακόλουθη ανάλυση που τότε είχα αναπτύξει. Συνήθως τέσσερις παράγοντες πρέπει να συνεπάρχουν ταυτόχρονα ώστε να ξεκινήσει μια πραγματική δημοκρατική μετάβαση σε μια πολιταρχική χώρα. Πρώτον, πρέπει να υπάρχει μια γενικευμένη δυσαρέσκεια από τον κοινό, από τους πολίτες. Δεύτερον, διέρεση στην ηγεσία του απολυταρχικού καθεστώτος. Τρίτον, δημοκρατική αντιπολίτευση και τέταρτον, διεθνής υποστήριξη. Όλα αυτά μαζί με μια μαγική συνταγή που ονομάζεται κρίση ήμουν σίγουρος ότι αυτή η κρίση θα έρθει και ότι θα ήταν είτε τεχνητή είτε φυσική. Λόγω της φύσης του καθεστώτος, η λαϊκή δημοκρατία όπως και η Σοβιετική Ένωση γνωρίζει τις στιγμές της του Τσερνομπίλ, λέει ο Μιλτής. Δεν μου επιτρέπει το χρονικό μου πλαίσιο να επεκταθώ πολύ περαιτέρω για την επιδημική κρίση, αλλά είμαι στη διάθεσή σας για ερωταπαντήσεις. Ως προς τη διεθνή στήριξη, ήθελα να υπογραμμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σίγουρα θα πρέπει, μάλλον πολύ σύντομα θα πρέπει να αναπτύξει ένα σχέδιο αντιμετώπισης της ε, μόχλευσης που ασκεί η Κίνα παγκοσμίω, χρησιμοποιώντας την καταστροφή αυτή και μάλιστα θυσιάζοντας την ζωή πολλών πολιτών της και τη ζωή πολλών ξένων υπηκόων. Ας ελπίσουμε όλες αυτές οι θυσίες να μην, είναι, να μην έχουν υπάρξει μάταιες. Έχω επίσης συστάσεις συγκεκριμένες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι στη διάθεσή σας να σας τις πω αν θέλετε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γιάνν Λιγιάνγκ. Έχουμε και την Σάρα Μπρούξ που θα μας μιλήσει για την Κίνα και μετά θα δώσω το λόγο στα μέλη για ερωτήσεις θα πρέπει να περιμένετε λίγο και μετά θα έχουμε την ώρα των ε, ερωταποκρίσεων. Η κυρία Μπρούξ, ε, σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε εδώ σήμερα. Η Διεθνής Υπηρεσία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι μια οργάνωση που τα τελευταία 35 χρόνια υποστηρίζει του υπέρμαχους ανθρωπίνων δικαιωμάτων έτσι ώστε η κοινωνία των πολιτών να χρησιμοποιήσει τα Ηνωμένα Έθνη για να προασπίσει τους πολίτες. Έτσι μπορούν να συνεισφέρουν στην ειρήνη, δικαιοσύνη, ισότητα και βιωσιμότητα. Αποτελούν αναπόσπαστο μέρος πολλών προσεγγίσεων των Ηνωμένων Εθνών. Παρά τις αδυναμίες του, το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών δημιουργεί δυνατότητα για αλλαγή. Έτσι η ομάδα μας υποστηρίζει όλους τους ακτιβιστές από την Νότιο Κορέα μέχρι την Γαλλική Ουιάννα, την Δυτική Αφρική και την Κεντρική Αφρική μέσω Ηνωμένων Εθνών. Επειδή μιλάμε επί αυτού του θέματος στο πάνελ, τα ολοκληρωτικά καθεστώτα είναι διαφορετικά. Όταν οι πολίτες δεν μπορούν να δράσουν και όταν τα δικαστήρια δεν ελέγχουν την εξουσία, τότε οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν ελάχιστες διόδους. Γι' αυτό αυτός ο πολυεπίπεδος χώρος είναι ύψης της σημασίας θα εστιάσω την προσοχή μου στη συμμετοχή, τον εκφοβισμό και νέα ερμηνεία του κανονιστικού πλαισίου. Μία από τις πιο ανησυχητικές τάσεις είναι ότι κλείνει ο χώρος παρέμβασης στα Ηνωμένα Έθνη. Αυτό το βλέπουμε και για οργανώσεις όπως η ΕΟΚΕ. Η Κίνα επίσης λογοκρίνει την γλώσσα που χρησιμοποιούν οι ΜΚΟ, ακόμα και στις ιστοσελίδες των ΜΚΟ. Και η Ινδία επίσης φημώνει οργανώσεις. Η δανέζικη οργάνωση International Dalit Solidarity ε, είδε ότι δεν μπορούσε να λάβει διαπιστευτήρια την τελευταία φορά που έδρασε. Γι' αυτό προσπαθήσαμε να ε, προωθήσουμε την, τις αρχές της διαφάνειας λογοδοσί, και λογοδοσίας κάτι το οποίο δεν ισχύει στην περίπτωση της Κίνας και της Ρωσίας. Βλέπουμε ότι όταν αποστέλλεται ηλεκτρονικό ταχυδρομείο υπάρχει φοβισμός και αντίπεινα από τις χώρες αυτές. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών από το 13 έως το 18 ανέφερε ότι η Κίνα είναι από τις χώρες που παραβιάζουν πολύ περισσότερο από άλλες. Αυτό αφορά εκφοβισμό, οχλήσεις, κρατήσεις και διώξεις. Το ίδιο διαπιστώνουμε και στην Αίγυπτο. Είδαμε ότι πολλά πρόσωπα που συμμετείχαν στο UPR το 2014 δεν μπορούν να βγουν από τη χώρα έξι χρόνια αργότερα και έχουν οδηγηθεί στη φυλακή για 25 χρόνια. Αυτό το βλέπουμε και σε άλλες χώρες που δεν λογοδοτούν. Επίσης, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η, η ανεξαρτησία των μέσων. Παρακαλούμε να μιλάτε λίγο πιο αργά. Αυτό που κάνουν αυτές οι κυβερνήσεις σαν στόχο είναι να φημώσουν τους επικριτές και δείχνουν ότι χρησιμοποιούν όχι μόνο τη δύναμη της πυθούς, αλλά και τη δύναμη του πορτοφολιού. Το 2018 ο πρέσβης της Κίνας ε, έκανε μία δήλωση στην ύπατη αρμοστία που ε, αναφέρθηκε σε γεγονότα τα οποία θεώρησε απαράδεκτα ως προς την κοινωνία των ε, πολιτών. Παράλληλα, ο ε, ύπατος εκπρόσωπος Ζαΐντ θεώρησε ότι θα πρέπει να τορπιλήσει την εργασία της ύπατης αρμοστίας. Έτσι, οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες έπρεπε να υποστούν τον εκφοβισμό που προβάλλουν αυτοί οι φορείς. Επίσης, αυτό αφορά και την Επιτροπή Προϋπολογισμού των Ηνωμένων Εθνών. Η Κίνα και η Ρωσία ε, ζητούν περιστολή και περιορισμό των κονδυλίων, ιδιαίτερα σε σχέση με την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Κίνα και η G77 θεώρησαν ότι θα πρέπει να μειωθούν τα κονδύλια υπεράσπισης της κοινωνίας των πολιτών. Το μέλλον της Διεθνούς ε, Αμερόληπτης Επιτροπής στη Συρία και το Μιανμάρ που είναι προτεραιότητες για μας ως προς τις παραβιάσεις, παραβιάσεις με ε, θεωρεί η Κίνα, η Ρωσία και το Μπουρούντι καθώς και το Ιράν ότι δεν δρούν σωστά και θα πρέπει να περισταλεί η δραστηριότητά τους. Οι οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών ε, δεν δρούν αποδοτικά. Αυτό δημιουργεί προκλήσεις για την κοινωνία των πολιτών και αυτό που έχει σημασία είναι αυτοί οι οργανισμοί να τύχουν υποστήριξης. Επίσης, ε, γίνεται νέα ερμηνεία ενιών που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το πρόγραμμα δράσης και η δήλωση της Βιέννης, ένα έγγραφο του 1993, τονίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι καθολικά και αδιέρετα. Το 2013 μέχρι 2015 η Ρωσία μίλησε για ε, παραδοσιακές αξίες και προστασία της ε, οικογένειας. Αυτό σήμαινε ότι προωθούνται ε, αρχές κατά τον ΛΟΑΔ. Πρόσφατα η κινέζικη κυβέρνηση έχει απαλείψει μια συγκεκριμένη ορολογία ιδιαίτερα των όρων υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επειδή λοιπόν υπάρχει και η δράση μίας διαπεριφερειακής ομάδας που υποστηρίζει την δήλωση της Βιέννης, βλέπουμε ότι αυτές οι προσπάθειες των δύο καθεστώτων απέτυχαν. Αυτή η πρωτοβουλία ασχολείται με συνεργασία ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έναν επικοδομητικό διάλογο που είναι στόχος αφεαυτού. Και τέλος, πώς τα Συμβούλια Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα πρέπει να επανισορροπηθούν μέσα στα πλαίσια της εντολής. Άρα εστιάζουμε την προσοχή μας σε τρεις τομείς. Ε, καταρχήν, τις προκλήσεις από τα απολυταρχικά κράτη που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ενισχύσει το χώρο της ε, κοινωνίας των πολιτών στα Ηνωμένα Έθνη και μιλήσει για τον καθολικό χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το σύστημα το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή μετά το 45 θα μπορέσει να αντισταθεί. Θα απαντήσω στη διάρκεια των ερωταποκρίσεων. Θα ήθελα να πω όμως ότι δεν θέλουμε να κρατήσουμε ένα σύστημα αυτό καθεαυτό προστατεύοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα υποστηρίζουμε τα Ηνωμένα Έθνη έτσι ώστε τα πολιταρχικά καθεστώτα να μην μπορούν να δράσουν και να βοηθήσουμε αυτούς που αντιστέχονται στα καθεστώτα αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα δίνω το λόγο στα μέλη η Ιζαμπέλ Βίσλερ καταρχήν από το ΕΛΚ. Ε, ευχαριστώ πολύ ε, λυπάμαι κύριε Βουλέ που δεν ήμουν παρούσα για να ακούσω τη δική σας ε, παρέμβαση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές για αυτά που άκουσα. Νομίζω ότι όλοι είμαστε πολύ ευαισθητοποιημένοι σε αυτά που θίξατε, γιατί αυτό που έχει σημασία είναι να μπορεί κανείς να εκφραστεί ελεύθερα. Όταν δούμε τι συνέβη με τον κορονοϊό, καταλαβαίνουμε ότι εάν είχε υπάρξει ελεύθερη έκφραση, θα είχαμε να κάνουμε με μία τελείως διαφορετική κατάσταση. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ε, λοιπόν να δούμε τι ολέθριες συνέπειες έχει η περιστολή του δικαιώματος έκφρασης. Μας υποσχεθήκατε ότι θα μας, μιλήσατε, ε, θα μας μιλήσετε για συστάσεις. Θα ήθελα να τις ακούσω. Γιατί μας είπατε ότι θα μας μιλήσετε για συγκεκριμένες δράσεις και ελπίζω να έχετε να μας πείτε πιο να μας δώσετε πιο σαφή στοιχεία. Μιλάτε για δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών, αλλά μας λέτε ότι είναι ένας τόπος που μας δίνει πολλές δυνατότητες. Ένας κοινό τόπος. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε τι βλέπετε σαν ε, δυνατότητα δράσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ιζαμπέλ Σάντος από τους Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Προς τον κύριο Γιάνν Λί θα ήθελα να πω ότι συμμερίζομαι τις ανησυχίες του για τον απόλυτο έλεγχο αυτού του συστήματος τύπου μεγάλου αδελφού που εντατικοποιείται και ε, συρρυκνώνει το δημόσιο χώρο ελεύθερης έκφρασης, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μειονότητες όπως οι Θιβετιανοί και οι Ουιγούροι. Μιλάμε λοιπόν και για μειονότητες αλλά και οργανώσεις ε, και ακτιβιστές. Δυστυχώς υπάρχει μεγάλη επαγρύπνηση, αλλά τα δικτατορικά καθεστώτα χρησιμοποιούν τα μέσα εποπτείας για εκφοβισμό και παρακολούθηση και βλέπουμε ότι αυτό προσπαθεί να κάνει και η Κίνα και δια της οικονομικής ε, οδού ε, μεταφέροντας τα καπιταλιστικά διδάγματα στην ε, τοπική κοινωνία. Σε σχέση με τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την παρέμβαση της κυρίας Μπρούξ, Πιστεύω ότι τα Ηνωμένα Έθνη είναι ένας βασικός χώρος δράσης, αλλά υπάρχουν και πολλές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που παραπονούνται για ολοένα και μεγαλύτερη δυσκολία πρόσβασης στο καθεστώς του παρατηρητή έτσι ώστε να εισακουστούν ή να άκουστούν από τα Ηνωμένα Έθνη. Θα ήθελα να μας πείτε τι θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ε, πολυεθνικό επίπεδο για να μπορέσει να εισακουστεί. Γιατί δεν υπάρχουν έχουν εύρωστες ε, δημοκρατίες χωρίς ε, εύρωστες ε, κοινωνίες των πολιτών που η φωνή των οποίων ακούγεται στις διάφορες οργανώσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. ID. Ευχαριστώ πολύ όλους τους ομιλητές. Ακούσαμε κάτι το πολύ σκόπιμο από την κυρία Μπρούξ, ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών στα Ηνωμένα Έθνη, γιατί ε, έχουμε πληθώρα συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ε, αυτή τη στιγμή απειλείται από την κινέζικη εξουσία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας εξηγήσατε τα βήματα που έχει κάνει η Κίνα προς αυτή την κατεύθυνση. Θα ήθελα να μου πείτε ποιες είναι οι υποδείξεις σας ως προς τη διάσκεψη κορυφής Κίνας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρείτε ότι θα έχει το θάρρος η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην μιλήσει για στρατηγική εταιρική σχέση, αλλά να αντιταχθεί στους Κινέζους σε σχέση με αυτή την ε, συστημική ε, καταστολή και πώς βλέπετε το σχέδιο αυτό μία ζώνη, ένας δρόμος πώς μπορεί να ε, ενταχθεί στην ευρωπαϊκή, στα ευρωπαϊκά δεδομένα, διότι η Κίνα έχει μεγάλα συμφέροντα στην Ευρώπη, το ξέρουμε αυτό. Και ξέρουμε ότι η Ευρώπη είναι διχασμένη και 17 κράτη-μέλη ε, έχουν οικονομικούς ε, δεσμούς ε, με την Κίνα. Ας δούμε το λιμάνι του Πειραιά της Ελλάδας που ανήκει στην Κίνα. Θα θέλαμε να μας πείτε κύριε Γιάνγκ πώς εσείς βλέπετε, πώς θα έπρεπε να αντιδράσει μάλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτή την τάση της Κίνας. Ως προς το Τσερνομπίλ στο οποίο αναφερθήκατε, πιστεύετε ότι επίκειται, επίκειται εκ νέου. Είπατε ότι δέκα χρόνια πριν ε, πιστεύαμε ότι δεν θα υπήρχαν μεγάλες αλλαγές τα επόμενα 2-3 χρόνια, αλλά τα επόμενα 10. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει, ποιες θα είναι οι αλλαγές στην Κίνα την επόμενη δεκαετία. Σας ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσω το λόγο στον καλεσμένο μας από την Κίνα, θα ήθελα να ξαναδούμε την στρατηγική Κίνας Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2019. Ε, έχω ορισμένες αμφιβολίες ως προς τους στόχους της Επιτροπής, ε, δηλαδή με βάση τα συμφέροντα και τις αρχές η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εμβαθύνει τις σχέσεις για να προωθήσουμε τα κοινά μας συμφέροντα σε διεθνές επίπεδο. Ποια είναι τα κοινά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας σε παγκόσμιο επίπεδο. Μετά από όλες αυτές τις μαρτυρίες ε, για την εσωτερική οργάνωση της Κίνας ως προς το δίκαιο και την ε, οργάνωση των κοινωνικών δομών στην Κίνα. Βλέπουμε ότι η Κίνα έπρεπε να συνεργαστεί στα πλαίσια των συμφωνιών του Παρισιού, για παράδειγμα αλλά η Κίνα είναι πραγματικά έτοιμη να δουλέψει με βάση ευρωπαϊκά πρότυπα είτε στον τομέα των κλιματικών αλλαγών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εμπορικών συναλλαγών ή θέλει να αλλάξει τα διεθνή πρότυπα έτσι ώστε η Ευρώπη να υποταχθεί στα κινέζικα πρότυπα. Ποιος είναι ο βαθμός ειλικρίνειας ε, σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας. Σας υποβάλλω το ερώτημα και στους τρεις γιατί συμμετέχετε στις εργασίες στα Ηνωμένα Έθνη και βλέπετε πώς εξελίσσονται τα πράγματα, άρα ίσως θα μπορούσατε να μας μιλήσετε για τους ειλικρινούς στόχους, αν υπάρχουν, της κινέζικης κυβέρνησης. Δίνω τον λόγο στον καλεσμένο μας από την Κίνα και μετά θα δώσω το λόγο στο, στην κυρία Μπρούξ και στον κύριο Βούλε. Ο κύριος Γιάνγκ έχει το λόγο. Έχετε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρίες και κύριοι για τις πολύ σημαντικές ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις είναι τόσο πολλές ώστε δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Θα ξεκινήσω με το σημαντικότερο νομίζω την επιδημία του ιού. Η κακή απόδοση ενός αυταρχικού συστήματος κρύβεται μέχρι να προκύψει κάποια κρίση, είτε οικονομική, είτε περιβαλλοντική, είτε πόλεμος, με διεθνής ταπείνωση ή ένα σκάνδαλο διαφόρας. Όταν συμβούν αυτά τα πράγματα, πλέον είναι προφανές ε, το τι συμβαίνει. Θεωρώ λοιπόν πως η τρέχουσα κρίση στην Κίνα είναι αυτή η στιγμή. Η επιδημία θυμίζει την καταστροφή του Τσερνομπίλ στην Σοβιετική Ένωση. Δεν είναι μια απλή παρομοίωση. Τα ίδια πράγματα συμβαίνουν στην Κίνα. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα που είχα χρησιμοποιήσει πριν από λίγα χρόνια σε μια άλλη ακρόαση. Ο πρώτος παράγων ο οποίος κοιτάμε είναι η γενική ικανοποίηση των ανθρώπων. Το καθεστώς αυτό λοιπόν ε, έχει εχθρούς, ε, αντιφρονούντες, ανεξάρτητους διανόμενους, ε, μειονότητες, ε, ανθρώπους στο Χονγκ Κόνγκ κτλ. Αλλά επειδή αυτή η επιδημία αποκάλυψε τις αδυναμίες του Καστοτός, θα ενταθεί η δυσαρέσκεια του κόσμου θα δημιουργήσει ε, οργή, ειδικά μετά τον θάνατο του γιατρού Λί. Μια ολόκληρη γενιά απαιτεί ελευθερία λόγου. Και τόσοι πολλοί διανοούμενοι, οι οποίοι συνήθως σιωπούν, ε, τώρα μιλάνε. Τότε βλέπουμε τη δυσαρέσκεια του λαού με την κυβέρνηση αυτή η οποία ενδύνεται. Και ενδύνεται και η απέτηση για αλλαγή. Τώρα. Ο πιο σημαντικός παράγοντας νομίζω είναι η οικοδόμηση μιας βιώσιμης δημοκρατικής αντιπολίτευσης Πολλοί όμως ε, διανοούμενοι μιλάνε για το θέμα αυτό. Και άρα υπάρχει εδώ πέρα ένας διχασμός εντός του καθεστώτος. Ξέρετε ότι μετά το ξέσπασμα της επιδημιάς ο Σιζιν Jinping για πρώτη φορά άφησε τον Πρωθυπουργό να προεδρεύσει της σχετικής ομάδας ε, της Επιτροπής που είχε αρμοδιότητα για την επιδημία και πήγε στο Βουχάν. Μία φορά μόνο. Μετά έχει σχεδόν εξαφανιστεί από τις ειδήσει. και το όνομά του δεν αναφέρεται πλέον. Και στην μικρή ομάδα στην οποία προεδρεύει δεν υπάρχουν στρατιωτικοί. Αυτό σημαίνει ότι ο Xi Jinping δεν τον αφήνει να διατάξει στρατό. Και κάποιοι ντόπιοι ε, εκφράστηκαν κατά του Xi Jinping και λένε ότι δεν φταίνε αυτοί για το χάλι στις αρχικές φάσεις, αλλά η ανώτατη ηγεσία που δεν τους επέτρεπε να ενημερώσει τον κόσμο. Οπότε η ανώτατη ηγεσία φταίει για τα χάλια αυτά και και πριν από λίγες μέρες το περιοδικό του κόμματος ε, δημοσίευσε ένα άρθρο ε, για την ομιλία του Xi Jinping που αποκάλυψε ότι ε, στις 7 Ιανουαρίου ο Xi Jinping ήξερε ήδη για την επιδημία αλλά από τις 7 Ιανουαρίου μέχρι τις 20 Ιανουαρίου όταν δημοσιοποιήθηκε στην Κίνα η υπόθεση ε, είναι δύο εβδομάδες και οπωσδήποτε υπεύθυνο είναι ο Jinping. Αλλά το ερώτημα είναι γιατί δημοσιεύτηκε αυτή τη στιγμή αυτό το άρθρο. Όλα αυτά μας δείχνουν πως ε, υπάρχουν κάποιες ρογμές στην ηγεσία και με την επικοινωνία που έχω με ανθρώπους εντός της κυβέρνησης ε, γίνεται μια προσπάθεια από πολλούς αξιωματούχους να ε, ξαναδούν ε, το πώς έχουν τα πράγματα. Τέταρτον, η διεθνής στήριξη. Νομίζω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταστρώσει σχέδια ανάγκης για να βοηθήσει την Κίνα να ε, διαμορφώσει το, τη μελλοντική τους αντίδραση και να υπάρχει ελευθερία λόγου για τον κινέζικο λαό. Αυτά προτείνω εγώ ως αντίδραση στο θέμα αυτό και έχω και κάποιες άλλες συστάσεις. Δεν ξέρω αν έχω χρόνο να τα πω. Για την ώρα θα δώσω λόγο στην κυρία Μπρουκ. Και αν έχω την ευκαιρία θα περάσουμε και σε άλλες ερωτήσεις. Ευχαριστώ κυρία Μπρουκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολλές ερωτήσεις οι οποίες μάλλον εμπίπτουν σε τρεις ε, κατηγορίες. Η μία αφορά στο γιατί ακόμα βλέπουμε πολλές οργανώσεις που θέλουν να συμμετάσχουν στο διάλογο με τη χώρα αυτή, μετά οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και, με, και μετά πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να υπερασπιστεί το σύστημα πολυμέρειας ώστε να προστατεύσει την ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Για την πρώτη κατηγορία. Ε, αντιλαμβάνομαι ότι ίσως είμαι υπερβολικά αισιόδοξη. Υπάρχουν πολλές οργανώσεις στον κόσμο που βλέπουν τον ΟΗΕ όχι ως ε, μαγική λύση, αλλά ως πλαίσιο για να υποβάλουν τις ιδέες και τις προτάσεις τους. Ζητούν παρεμβάσεις στο Συμβούλιο, αλλά αυτά τα χρησιμοποιούν εσωτερικά στις χώρες τους, ώστε να συζητείτε το θέμα και να σκέπτονται λύσεις και δεν είναι εύκολα τα περιβάλλοντα αν σκεφτεί κανεί στην Κολομβία ή τις Φιλιππίνες ή την ακτή ελεφαντοστού αλλά πολύ συχνά σημαντικό τμήμα άλλων αυτών και ως προς την πρόσβαση των μη καπαόμικρων. Είναι σαφές ότι η κοινότητα των μη καπαόμικρων στη Νέα Υόρκη ε, δρά ως θεματοφύλακας παρά ως διευκολυντής ώστε να έχουν βήμα, να έχουν λόγο στα Ηνωμένα Έθνη. ώστε να υπογραμμίζεται ο σημαντικός ρόλος της κοινωνίας των πολιτών. Πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες, αλλά και στο επίπεδο του καθεστώτος μέλους και οι ευρωπαϊκές οργανώσεις μη καπάω μικρών να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αυτή χρειαζόμαστε βιώσιμη χρηματοδότηση για το σύστημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ και αντιμετώπιση αυτής της τάσης μείωσης χρηματοδότησης για τους εμπειρογνώμονες που παρακολουθούν τα θέματα αυτά. Μαζί με άλλες προσπάθειες που προσπαθούν να ενισχύσουν το πλαίσιο αυτό των Ηνωμένων Εθνών, όχι μόνο για να αντιμετωπίσουμε το έλλειμμα αξιοπιστίας, αλλά και για να αντιμετωπίσουμε άλλες δυνάμεις που θέλουν, προσπαθούν να κερδίσουν το πάνω χέρι. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2019 για τις προτεραιότητες των Εθνών και τις χθεσινοβραδινές στην ουσία πρέπει να αυξάνεται το πολιτικό κόστος και οικονομικό κόστος για τις κυβερνήσεις που προχωρούν σε καταπίεση του πληθυσμού για παράδειγμα μια υπερασπίστρια των ε, δικαιωμάτων των γυναικών στην Κίνα η οποία έχασε τη ζωή της, Αχμέτ Μανσούρ, που είναι φυλακισμένος επειδή ε, ε, έστελνε πληροφορίες στα Ηνωμένα Έθνη, στη Σαουδική Αραβία, που πληρώνουν υψηλό το τίμημα για την υποστήριξη αντίστοιχη ακτιβίστριας από την Κίνα. Οι χώρες του Μπενελούξ και η Γερμανία έχουν φέρει συγκεκριμένες περιπτώσεις ενώπιον του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών. Πρέπει να συνεχιστεί αυτή η πίεση ώστε να υφίσταται κόστος για τις κυβερνήσεις αυτές να αποτρέπουν την κοινωνία των πολιτών τους να συμμετέχει στα Ηνωμένα Έθνη για τα κοινά συμφέροντα σκεπτόμενοι κάπως το πλαίσιο των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας μαζί με τη Human Rights Watch, το, την Εκστατεία, το Θιβέτ, έχουμε συνεργαστεί και πολλές άλλες οργανώσεις, έχουμε συνεργαστεί την τελευταία δεκαετία με τον ΙΕΒ για τις προσδοκίες για τον διάλογο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πώς ο διάλογος αυτός τροφοδοτεί και την σύνοδο κορυφής με την Κίνα. Πολλοί από εμά στην αίθουσα θα συμφωνούσαν ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν είδαμε να μοχλεύεται ο διάλογος ώστε να αλλάξει η συζήτηση στα υψηλότερα επίπεδα ηγεσία για τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ως προς την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα επικεντρωνόμουν στο λεγόμενο 17 1 που είναι υψηλή ανησυχία αλλά βλέπουμε κάποιες διαρροές η Τσεχία είχε ήδη πει ότι δεν θα συμμετάσχει στο 17 συν 1 κάποιες πιέσεις από τα βαλτικά κράτη για την υπεράσπιση των ευρωπαϊκών αξιών και ε, ώστε να μην γίνονται αυτές οι χώρες ε, υποχείρια άλλων. Στον ΟΗΕ έχουμε δει βέβαια τι συμβαίνει όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, ομιλεί με ενιαία φωνή. Ιδιαίτερα όταν απέτυχε το 2017 η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει ενιαία δήλωση υπό το κεφαλαίο 4, δηλαδή δεν περιορίζεται στην Κίνα, θα μπορούσα να μιλήσω και για την κλιματική αλλαγή, αλλά είμαστε σίγουροι ότι δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολλά και διάφορα επίπεδα μπορεί να δράσει τον ΟΗΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε, θα ήταν σε θέση να οικοδομήσει μια αποτελεσματική στρατηγική για να αντιμετωπίσει τις απολυτερικές κυβερνήσεις σχετικά με το παρελθόν τους και να διευκολύνει το σύστημα λογοδοσίας ε, του, του πλαισίου υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διεθνώς, θα μπορούσε να καταρτήσει μια στρατηγική και να εντοπίσει δεσμεύσεις ώστε να υπάρξει ένας κανόνας, ένα πλαίσιο κανόνων λογοδοσίας που να είναι και υλοποιήσιμη στο έδαφος, στο πεδίο θα μπορούσε να δουλέψει πολύ καλύτερα με τα κράτη-μέλη ώστε να είναι εγγυητής όχι μόνο των δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά πολλών άλλων σχετιζόμενων ζητημάτων και ιδιαίτερα εσωτερικών που έχουν άμεση επίπτωση στην αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ομιλεί ως υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εξωτερικό. Και για να κλείσω, Νομίζω ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου είναι σαφή. Και εν συντομία, η Ένωση και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υπρασπιστούν ένα ισχυρό σύστημα των ΗΕ με βάση τα συμπεράσματα. Είναι υπέρ της αποτροπή των παραβιάσεων και της αντιμετώπισης τους. Ο ΙΕ έχει τρεις πυλώνες, ειρήνη, ασφάλεια και ανθρώπινα δικαιώματα στο μείγμα αποδυναμώνεται ο πυλώνας των δικαιωμάτων και αυτό απειλεί με κατάρρευση του όλου οικοδομήματος. Δεν θα μιλήσω για τις χώρες αυτές που μας απασχολούν τώρα, όπως για την Κίνα, γιατί θα πρέπει να προωθήσουμε διάλογο με τις εμπλεκόμενες χώρες. Ζήτησα να επισκεφθώ την Κίνα. Ελπίζω να μου δοθεί η άδεια και θα προωθήσω μία ε, ανάλυση, θα κάνω μία ανάλυση. Θα ήθελα όμως να μιλήσω για τις πιέσεις ε, κατά του ε, συστήματος διεθνών σχέσεων. Το διεθνές σύστημα είναι και το πλέον προσήκον και σε αυτό προστρέχουν τα θύματα. Μερικά όμως κράτη οργανώνονται για να ε, εξαφανιστεί αυτό το σύστημα, το οποίο δείχνει ότι το σύστημα ακούει τα θύματα. Θα ήθελα να πω σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί δύναμη παρόλο που ακούμε τη φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολλά ε, επίπεδα και φόρα, αλλά θα πρέπει να, ε, ε, να ακούγεται και σε περιφερειακούς φορείς. Ως προς αυτή την πίεση προς το διεθνές σύστημα, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποθαρρύνει αυτά τα κράτη-μέλη να συγκλίνουν προς ψηφίσματα τα οποία ενισχύουν το σύστημα, έτσι πιστεύουν, αλλά στην ουσία αποδυναμώνουν το σύστημα. Θα πρέπει να αποθαρρύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση κράτη να υποστηρίζουν αυτά, τέτοια ψηφίσματα. Επίσης, θα πρέπει να γίνει μια συμμαχία με τις χώρες του Νότου, γιατί οι χώρες οι οποίες θέλουν να αποδυναμώσουν το διεθνές σύστημα είναι οι χώρες που προέρχονται από το Νότο. Θα πρέπει λοιπόν να υποθεί σε αυτές τις χώρες του Νότου ότι όταν μιλάμε για την ε, κοινωνία των πολιτών σημαίνει, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μία επιμερισμένη ανάπτυξη και δεν θα πρέπει να εντάξουμε αυτές τις χώρες σε πρωτοβουλίες οι οποίες είναι επιζήμιες προς το διεθνές σύστημα. Θα πρέπει να κινηθούμε πέρα λοιπόν από το σύστημα. θεωρούμε ότι υπάρχει επαρκής κατανόηση του ζητήματος. Όταν υφίσταται ένα ζήτημα θα πρέπει να το αναλύει η διεθνής κοινότητα και τα θύματα πρέπει πάντα να τυχαίνουν προστασίας. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να ε, ε, έχει το λόγο, να έχουν το λόγο οι οικονομικές δυνάμεις, αλλά και οι πολιτικοί που έχουν τα ίδια συμφέροντα με τους πολίτες. Ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε στη Ρωσία. Δίνω το λόγο στην ε, κυρία Λασίλα που είναι υπεύθυνη του Φιλανδικού Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων θα μας μιλήσει για τη Ρωσία και τις πρόσφατες εξελίξεις, τη συνταγματική αναθεώρηση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Υποεκτροπής των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θα μιλήσω για δύο πτυχές ε, της ε, τρέχουσας ε, συνταγματικής μεταρρύθμισης. Υπάρχει η ομιλία του πρόεδρου Πούτιν στις 15 Ιανουαρίου για την επίσημη εκκίνηση του ούτως αποκαλούμενου προβλήματος του 24 όταν δηλαδή ολοκληρώνεται η θητεία η δεύτερη θητεία συνεχιζόμενη αυτή τη φορά του πρόεδρου Πούτιν. Επίσης η ανταπόκριση του καθεστώτος λέει ο ομιλητής απέναντι σε μια όλο και πιο ανήσυχη κοινωνία των πολιτών τα οποία έχουν γίνει μεγάλος πονοκέφαλος για το Κρεμλίνο. Ο Βλαδίμρος Πούτιν ε, ανακοίνωσε συνταγματικές ε, τροποποίησεις και θεωρείται πλέον ε, σταθμός στην ανάπτυξη του ρωσικού απολυτερχικού στήματος το τρέχον σύνταγμα του 1993 βασίζεται σε φιλελεύθερους στόχους και ευθυγραμμίζεται με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ρωσίας. Οι προβλεπόμενες αλλαγές θα έχουν σχέση με το διεθνές δίκαιο. Αντί να ευθυγραμμίζεται το Σύνταγμα με το διεθνές δίκαιο, πλέον θα ευθυγραμμίζεται μόνο με το σώμα του ρωσικού δικαίου σημαντικό ζήτημα υπό τη σκοπιά αυτή είναι η μελλοντική στάση της Ρωσίας ε, ή η συμμόρφωσή της προς τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και ε, αποστέλει ένα πολιτικό μήνυμα προς όλους τους διεθνείς παίκτες. Δηλαδή η Ρωσία θέλει να αποδείξει στους ε, εξένους ότι δεν έχει κανένα νόημα να της ασκείται πίεση επί τη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι δύσκολο να πει κανείς αν αυτό θα σηματοδοτήσει την μεταφορά από το παρόν σε ένα μελλοντικό πρότυπο απολυταρχίας. Βέβαια αυτές οι αλλαγές ήδη από το 12 είχαν προανακοινωθεί όταν ξεκίνησε η τρίτη προεδρική θητεία στην ουσία του Πρόεδρου Πούτιν από την άλλη είναι λογικό να αναρωτηθεί κανεί κατά πόσον θα είχαμε δει τις εξελίξεις του, του Ιανουαρίου, αυτού του Ιανουαρίου, αν ε, είχαν ήδη αρθεί οι περιορισμοί των ε, δύο διαδοχικών ε, θητιών. Έχουμε πολυάριθμες παραβιάσεις των εγγυημένων ε, ελευθεριών της κοινωνίας των πολιτών από την κυβέρνηση, από το καθεστώς που την λέει ο μιλτής, και είναι σύμφωνα με τον νόμο ο πρόεδρος που καθορίζει, που ορίζει τι είναι οι ελευθερίες οι κοινωνικές μεταξύ άλλων. Φαίνεται ότι στο μέλλον θα είναι πιο μετριασμένες οι εξουσίες του Προέδρου όχι με το Κοινοβούλιο, αλλά με ένα νέο κρατικό φορέα που θα καθορίσει το νέο σύνταγμα. Αυτός ο φορέας μάλλον θα είναι το επί του παρόντος άτυπο κρατικό συμβούλιο. Και μάλλον την εξουσία του οργάνου αυτού θα αναλάβει ο ίδιος ο Πούτιν. ώστε να διαχυθούν οι σημερινές ε, γραμμές διακυβέρνησης του Πούτιν και η κατακόρυφη γραμμή εξουσίας που ακολουθεί. Όποιες άλλες αλλαγές και να φέρει αυτή η συνταγματική μεταρρύθμιση, η άλλη πτυχή που την αφορά το ζήτημα είναι η ρωσική κοινωνία που είναι όλο και πιο απογοητευμένη. Μέχρι το 2017, το αργότερο, η ούτως αποκαλούμενη ε, συνένεση της Κρυμαίας ε, είχε απαξιωθεί στα μάτια της κοινωνίας. Το 2017 για πρώτη φορά, κατά τη διάρκεια διακυβέρνησης Πούτιν, περίμεναν οι πολίτες μεγάλης κλίμακας ε, κοινωνικές αλλαγές, κατά άνω του 50%. Αυτή τη στιγμή, άνω του 60% της ρωσικής ε, κοινή νόμης αναμένουν απτές αλλαγές από την κυβέρνηση. Μέχρι στιγμής, ανέλαβε την κοινωνική πρωτοβουλία υπό τις ανακοινώσεις του Πούτιν το Κρεμλίνο, απομακρύνοντας την προσοχή από τα παρόντα έντονα ε, κοινωνικά προβλήματα προς προβολές και θεωρίες σχετικά με το μέλλον της συνταγματικής μεταρρύθμισης. Παράλληλα, το Κρεμλίνο προσπαθεί να ανταποκριθεί στις ε, αυξανόμενες απαιτήσεις για κοινωνική δικαιοσύνη. Πολύ πιο προβληματική είναι η δικαιολόγηση του πολιτικού συστήματος όταν υπάρχει στάση και υποχώρηση στην οικονομία, ε, λέει ο μιλτής, ε, και υπό την προπαγάνδα που εκπέμπει η κρατική τηλεόραση. Το 17 και 18 παρά την προπαγάνδα αυτή το ποστό των πολιτών που ήθελε να βασίζεται η ρωσική κοινωνία ε, σε φιλελεύθερες αξίες πιο κοντινές στη Δύση αυξήθηκε από 27% σε 37%. Αντίστοιχα, οι αξίες που ε, υποστήριζε το Κρεμλίνο υποχώρησαν, λέει ο μιλητής, από 35% σε 27%. Πάντω η εικόνα του Κρεμλίνου καταραίει και αυτό είναι το βασικότερό του πρόβλημα. Το καθεστώς ε, είναι όλο και πιο εξαρτώμενο από ε, πολιτικές καταπίεσεις και περιορισμού της ελευθερίας, η ιδιωτικοποίηση Ε, επιλεγμένων, ε, επιλεγμένου πελατειακού καταλόγου και η εστίαση σε συγκεκριμένα εξωτερικά θέματα χάνει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον του ε, για την ρωσική κοινή γνώμη. Η καταπίεση αυτή είναι πολύ πιθανό να συνεχιστεί. Έχει αναπτυχθεί νομοθεσία κατά των ξένων πρακτόρων, περιορισμοί για το διαδίκτυο, για τις μεταφορές χρημάτων πιο αυστηρές ποινές για συναθρήσεις που δεν έχουν ε, πάρει έγκριση. Επίσης, η αποδυνάμωση του, της δικαιοσύνης ε, έχει συνεισφέρει και αυτή. Οι αποφάσεις των δικαστηρίων ε, αποσκοπούν στο να αποδείξουν την ε, πίστη τους και την αφοσίωσή τους στο καθεστώς παρά την υπηρεσία τους στον νόμο η όλη δικαστική διαδικασία ε, ακολουθεί τις επιταγές του καθεστώτος. Λαμβάνει η χώρα βία και βασανιστήρια στις φυλακές, αυτό έχει αναγνωριστεί. Η δημοσιοποίηση περιπτώσεων βασανιστήριων σε τελευταία χρόνια αποτυπώνει ε, το γεγονός ότι επιβιώνει η κοινωνία των πολιτών και οι φωνές που διαφωνούν παρά το σύστημα το πολιταρχικό. Βεβαίως υπάρχει νομοθεσία που απαγορεύει, απαγορεύει οποιαδήποτε δραστηριότητα θεωρείται αντικρατική από τις αρχές. Το 19 είδαμε όμως μια νέα έκφραση αλληλεγγύης η περίπτωση του δημοσιογράφου Ιβάν Γκολούνοφ τον Ιούνιο του 19 ήταν σημείο καμπής όταν αποσύρθηκε η ε, δίωξη που του είχε ασκηθεί, μετά τις πολυάριθμες ε, συλλήψεις του καλοκαιριού του 19, είδαμε διάφορες ομάδες επαγγελματιών, ηθοποιών, δικηγόρων, ιατρών και άλλων, που πίεσαν να αποσυρθούν τέτοιες κατηγορίες και διώξεις. Ε, τέλος, η αλλαγή του συντάγματος προς πιο πολιτορχικές ε, κατευθύνσεις έχει καταστεί ιδιαίτερη ανησυχία για πολλές γενναίες ε, φιλελεύθερων ανθρώπων στη Ρωσία. Το Σύνταγμα του 1993 ήταν σημαντικό σημείο αναφοράς για την νομιμότητα διαφόρων κυβερνητικών πολιτικών και δράσεων. Παρόλα αυτά, το καθεστώς Πούτιν, και εδώ διακόπτεται η σύνδεση με τον ομιλητή. Okay. We are going to give the... Η Πρόεδρος. Θα δώσουμε τον λόγο στην κυρία Ράποβα από το Mass Media Defense Center της Ρωσίας και θα επανέλθουμε με τη σύνδεση του ομιλητή για τις ερωταπαντήσεις. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ε, good afternoon, ε, ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Ναι, συγγνώμη. Α, επανήλθατε. Ναι, ναι, υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα τα οποία όμως εξακολουθούν να υπάρχουν. Θα επανέλθουμε μετά για τις ερωτήσεις λοιπόν, λέει η πρόεδρος. Ωραία. Ε, το ίντερνετ μας δυσκολεύει. Ευχαριστώ που με προσκαλέσατε να μιλήσω για την ελευθερία έκφραση στην ε, Ρωσία. Θα ξεκινήσω με μια γενική παρουσίαση της κατάστασης όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης ε, και ΜΜΕ και θα σας δώσω κάποια παραδείγματα για το πόσο το νομικό πλαίσιο ε, δίνει κάποια μέσα στην κυβέρνηση για να ελέγξει την διάδοση πληροφοριών και την ελευθερία έκφρασης και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε σχετικά. Λοιπόν, γενικά η ελευθερία έκφρασης στη Ρωσία μειώνεται τα τελευταία 10-15 χρόνια Ε, στο διάστημα αυτό έχουν υπάρξει 13 διαφορετικά νομοθετήματα σχετικά που δίνουν τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να ελέγχει την ελεύθερη έκφραση το διαδίκτυο, την ροή πληροφοριών και να δίνει κάποια επιπλέον εργαλεία παρακολούθησης. Νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες οι οποίες περιορίζουν την ελευθερία έκφρασης και διαδικτύου έχουν στόχο να ενισχύσουν την τον έλεγχο της κυβέρνησης. Και πολύ πρόσφατοι νόμοι έχουν εγκριθεί με τη δικαιολογία της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού και όπως εξηγεί η ρωσική κυβέρνηση, τα μέτρα αυτά είναι απολύτως απαραίτητα και παρόμοια μέτρα ήδη ε, υπάρχουν και σε άλλες δημοκρατικές ε, ευρωπαϊκές χώρες ένα παράδειγμα, παραδείγματος χάρη, είναι οι νόμοι περιβλασιμίας και προστασίας δεδομένων. Κάποια από τα βασικά θέματα ήταν η επαναπινικοποίηση της παραπληροφόρησης, η εισαγωγή πολύ αυστηρών κανόνων για την προστασία προσωπικών δεδομένων, απαγόρευση της ανωνυμίας στο διαδίκτυο, αυξημένη επιτήρηση που υπονόμευσε και την ερευνητική δημοσιογραφία. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα εξοδικαστικού μπλοκαρίσματος ε, ιστοσελίδων με αποτέλεσμα να κλείνουν διάφορα ανεξάρτητα μέσα στο διαδίκτυο Και βεβαίως η έλλειψη ανεξάρτητου δικαστικού συστήματος σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο έω άσκοπο να προσφύγουμε στα δικαστήρια. Για καμιά φορά και επικίνδυνο. Οπότε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε πολλές περιπτώσεις είναι η τελευταία ελπίδα για τους Ρώσους δημοσιογράφους και ακτιβιστές να έχουν μια δίκαιη δίκη. Υπό αυτές τις συνθήκες ε, η δημοσιογραφία ανήκει στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα στην Ρωσία. Σύμφωνα με τους ε, δημοσιογράφους χωρίς σύνορα, το 2019 η Ρωσία βρίσκεται στη θέση 149 παγκοσμίω από 180 χώρες όσον αφορά την ελευθερία των ΜΜΕ. Και εδώ είναι τα βασικά ζητήματα. Όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης ε, και την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Ανέφερα ήδη ότι αποποινικοποιήθηκε η συκοφαντία το 2012, αλλά 12 μήνες μετά, 6 μήνες μετά, με συγχωρείτε, Και παρά το ότι βεβαίως δεν υπάρχει πλέον η ποινή της υπάρχουν τεράστια πρόστιμα. Κάτι το οποίο προκαλεί μια αυτολογοκρισία. Επίσης υπάρχει κατάχρηση της νομοθεσίας κατά του εξτρεμισμού. Χρησιμοποιούνται αυτές οι ποινικέ διατάξεις για να σοπάσουν οι επικριτές στο διαδίκτυο. Παραδείγματος χάρη, το 2017 95% των καταδικών αφορούσαν ε, ε, εκφράσει στο διαδικτύο και ήταν, ε, κειμενόταν από φυλακίσεις μέχρι καταναγκαστικά έργα και καταναγκαστική ιατρική θεραπεία. Άλλοι ειδικά τιμωρήθηκαν για το ότι εξέφρασαν αντιρρήσεις για την παρέμβαση στην Ουκρανία. Επίσης η βλασφημία ε, και οι σχετικοί νόμοι χρησιμοποιούνται ιδιαίτερως ε, ειδικά για όσους ε, εκφράζονται κατά της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και για τους blogger που χρησιμοποιούν εικόνες στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιήθηκε αυτή η διάταξη παραδείγματος χάρη πρόσφατα 17 φορές τα τελευταία χρόνια. Το δικαίωμα στη λύθη. Ο νόμος ο οποίος εισήχθη στην Ευρώπη. Έχει πολλά και διάφορα αφηρημένα πράγματα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι αρχές ε, για να απαγορεύσουν κάποιες δημοσιεύσεις ε, στο διαδίκτυο. Ειδικά όταν ασκούν κριτική σε αξιωματούχους. Οπότε έχουν αρκετά αποτελεσματικά μέσα για να αφαιρέσουν υλικό από το διαδίκτυο όταν αναφέρεται η διαφθορά τους. Ένα άλλο θέμα το οποίο έφερε η κυρία Μπρούξ ήδη είναι η ΛΟΑΤΚΙ και τα σχετικά ζητήματα. Η Ρωσία εισήγαγε το νόμο περί ομοφιλόφιλης προπαγάνδας ε, που δίνει την δυνατότητα δίωξης ε, ή ουδήποτε καλύπτει τέτοιες δραστηριότητες και οι διατάξεις αυτές ε, παρέχουν μέσα στις αρχές για να στιγματίζουν τους ΛΟΑΤΚΙ και εμποδίζουν και την πληροφόρηση για υγεία και εκπαίδευση. Ένα άλλο θέμα ο έλεγχος των κρατικών ΜΜΕ δηλαδή είτε είναι κρατικά τα κανάλια είτε ανήκουν σε κάποιους ε, κοντινούς. Ε, κάποια μημία αναγκαστικά να μετακομίσουν στο εξωτερικό για να βρουν ανεξάρτητη στήριξη και να μην υφίστανται έλεγχο από τις ρωσικές αρχές όπως ε, το Μεντούζα, ε, το Ντόστ και το σταθμός 2, τοπικό σταθμός στο Τόμσκ της Σιβηρίας που έχασε την αδειά τους, έχασαν την αδειά τους και εκπέμπουν στο διαδίκτυο. Αυτές είναι οι μόνες ε, πληροφορίες ε, που είναι διαθέσιμες ε, στο διαδίκτυο. Και είναι ακόμα ανεξάρτητες. Ένας άλλος τομέας είναι ο περιορισμός της ξένης ιδιοκτησίας απαγορεύεται σε ξένους υπηκόους και σε άτομα με διπλή υπηκότητα να ιδρύουν ε, είτε να είναι αρχισυντάκτες σε ρωσικά μιμιέ. Έτσι, υπάρχει λιγότερο πλουραλισμός και περιορίζεται η ελευθερία πληροφόρησης. Επίσης θα έχετε ακούσει ε, τον νόμο περί ξένων ε, πρακτόρων που χρησιμοποιείται κατά τον ΜΚΙΟ. Εγώ, ας πούμε, είμαι επικεφαλής ε, μιας ΜΚΙΟ που ασχολείται με την ελευθερία της έκφρασης. Οπότε και η δική μας η ΜΚΙΟ θεωρήθηκε ε, ξένο όργανο. Λοιπόν, τώρα ο νόμος αυτός θα χρησιμοποιηθεί κατά των ξένων ΜΜΕ και ατόμων ακόμα. Ε, οπότε ε, και αυτή την ανισχία θα ήθελα να ακούσετε. Γιατί βεβαίως ε, αναμένουμε να στραφεί αυτό κατά των επικριτικών φωνών και του πλουραλισμού. Τον Δεκέμβριο του 2019 τροποποιήθηκε ο νόμος περί ΜΜΕ ε, χωρίς διαβούλευση ε, και πλέον και άτομα μπορούν να θεωρηθούν ξένοι πράκτορες οποιοδήποτε ανεξαρτήτως υπηκότητας όποιος έχει εισόδημα στο εξωτερικό και ε, όσοι, όσοι είναι ανταποκριτές ξένων μιμιέ Οπότε αυτό ισχύει για δημοσιογράφους, blogger, επαγγελματίε, επαγγελματίες, ε, ακόμα και εμπειρογνώμονες ε, που εκφέρουν άποψη για ζητήματα. Αυτά λοιπόν ε, ετέθησαν εν ισχύ πέρσι. Τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει για να στοχεύσουν άτομα ως ξένους ε, πράκτορες αλλά είναι σαφής οι επιπτώσεις ε, του νόμου αυτού. Θα υπάρξει μια αυτολογοκρισία θα ασκηθεί πίεση σε ανεξάρτητους δημοσιογράφους να μην συνεργάζονται με ξένα ΜΜΕ να μην ε, μοιράζονται πληροφορίες ε, στο διαδίκτυο, ειδικά από ξένα ΜΜΕ, τα οποία θεωρούνται ήδη πράκτερες, όπως η Φωνή της Αμερικής, το Radio Liberty. και την παρουσία του στο διαδίκτυο. Οπότε έχουμε εδώ πέρα απειλή για την ελευθερία του λόγου στο διαδικτύο. Όσον αφορά τους περιορισμούς στο διαδικτύο. Λοιπόν, ε, όπως είπα ήδη, η Ρωσία έχει ένα νόμο που της δίνει τη δυνατότητα να μπλοκάρει διάφορα site χωρίς κάποια δικαστική απόφαση. Οπότε υπάρχουν έτσι οι δυνατότητες να μπλοκαριστεί το οτιδήποτε στο διαδίκτυο αυθαίρετα. Και δεν επιτυγχάνουν οι προσπάθειές μας στα δικαστήρια αρκετές ε, περιπτώσεις εκκρεμούν στο ΕΔΑΔ όπως ε, παραδείγματο χάρη το granny.ru, το Daily Journal και ε, τους εκπροσωπούμε τη συγκεκριμένη εφημερίδα ενώπιον του ΕΔΑΔ. Επίσης υπάρχει ο νόμος που αφορά την εξατομίκευση δεδομένων. Απαγορεύτηκε το LinkedIn στη Ρωσία γιατί ε, έπρεπε να δώσει τα στοιχεία των Ρώσων χρηστών στις ρωσικές αρχές. Ήδη λοιπόν έχει μπλοκαριστεί εδώ και 3,5 χρόνια. Τώρα αντιμετωπίζουμε μια παρόμοια κατάσταση με το Facebook και το Twitter που μόλις ε, ε, δέχτηκαν ένα πρόστιμο γιατί δεν συμμορφώνονται με τον νόμο αυτόν. 60.000 ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα. Και αν ε, δεν συμμορφωθούν, αν δεν πληρώσουν δηλαδή, ε, δεν θα υπάρξει απαλλαγή από την ανάγκη συμμόρφωσης. Δηλαδή, εντάξει, το Facebook είναι αρκετά δημοφιλές ε, στη Ρωσία, ειδικά για την αντιπολίτευση, την κοινωνία των πολιτών κτλ. Οπότε αν μπλοκάρει αυτή η πλατφόρμα ε, θα υπάρχουν αρνητικές συνέπειες στην ελευθερία της πληροφόρησης, ειδικά για την κοινωνία των πολιτών. Το τεράστιο πακέτο Γεραβάη, Γεραβάη είναι ο βουλευτής, ο οποίος είχε φέρει την ομοθεσία αυτή. Το πακέτο Γεραβάη λοιπόν ε, δικαιολογήθηκε ως αντιτρομοκρατικό. Και ήταν πάρα πολύ αρνητικό για το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, ελευθερία έκφραση κτλ. Και δίνεται η δυνατότητα στην κυβέρνηση να έχει όχι μόνο μεταδεδομένα ε, από τους παρόχους, αλλά και το περιεχόμενο. Τώρα λοιπόν οι πάροχοι είναι υποχρεωμένοι να καταγράφουν και να αποθηκεύουν όλες τις επικοινωνίες ε, ή ουδήποτε είναι στη ρωσική επικράτεια, όχι μόνο των Ρώσων πολιτών. Αν επισκεφτείτε π.χ. εσείς στη Ρωσία, ε, ο νόμος ισχύει και για εσάς. Οπότε όλα αυτά θα καταγράφονται για έξι μήνες το περιεχόμενο και τα μεταδεδομένα για τρία χρόνια. Οι πληροφορίε αυτές θα πηγαίνουν στις μυστικές υπηρεσίες χωρίς ε, δικαστικό έλεγχο. Αυτό βέβαια παραβιάζει την ιδιωτικότητα και την ελεύθερη διακίνηση πληροφοριών και την ελεύθερη έκφραση. Τώρα δεν θα αναφερθώ στην νομοθεσία που ασχολείται με αυτούς που συγκεντρώνουν τις ειδήσει ή τις μηχανές αναζήτησης και θα ήθελα να αναφέρω τρεις νόμους που πέρασαν πέρσι και είναι πάρα πολύ σημαντικοί ε, για το θέμα το οποίο μας απασχολεί σήμερα. Το ένα αφορά την ασέβεια προς αρχές, ε, το άλλο τους ευδείς ειδήσει. Ε. Και, και, και τα τρία πέρασαν επίσης χωρίς διαβούλευση. Το πρώτο προβλέπει και πρόστιμα για όσους διαδίδουν ειδήσει ε, που προσβάλλουν το Σύνταγμα, τις αρχές και τα σύμβολα του κράτους. Οπότε, ε, δεν μιλάμε για άνθρωπο δηλαδή ο οποίος προσβάλλεται ή θίγεται. Έχει χρησιμοποιηθεί ήδη 50 φορές κατά το τελευταίο έτος η συντηρητική πλειοψηφία των υποθέσεων ήταν ε, ε, δημοσιεύσεις ε, επικριτικές κατά του πρόεδρου Πούτιν ως αξιωματούχου. Τέλος. Οι δημοσιογράφοι στη Ρωσία υφίστανται εκφοβισμούς, κρατούνται σε διαδηλώσεις, απειλούνται, κατηγορούνται για διάφορα εγκλήματα δεν σχετίζονται απαραίτητο με τη δουλειά τους, αλλά ο λόγος είναι η επαγγελματική τους δραστηριότητα. Και θα ήθελα εδώ να αναφέρω τον Γκυρίδ ο οποίος είναι στο Καύκασος Νέτ ε, και ο οποίος καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση για κατοχή ναρκωτικών. Ένας άλλος συνάδελφος ε, για τον ίδιο λόγο απελευθερώθηκε μόνο με τα την παρέμβαση ε, άλλων δημοσιογράφων. Ένας άλλος δημοσιογράφος που πέρασε πάνω από 1,5 χρόνο κρατούμενος είναι ο Ιγκόρ Ρούντνικοφ, αρχισυντάκτης ε, των ανεξάρτητων ΜΜΕ του Καλίνιγκραντ. Ε, όπως είπα, 1,5 χρόνο πέρασε κρατούμενος και αφέθηκε ελευθερός χάρη στους δικηγόρους μας, οι οποίοι τον υπερασπίστηκαν ε, βρέθηκε στο στόχαστρο επειδή αποκάλυψε την διαφθορά τοπικών ε, ε, αξιωματούχων. Ένας άλλος δημοσιογράφος από το Νταγκεστάν, ο Μουμίρ Γκαρτζίεφ, κρατείται ακόμα για χρηματοδότηση της νομοκρατίας. Και Μία από τις χειρότερες περιπτώσεις αφορά την κυρία Προκόπιεβα, ε, η οποία εργάζεται για τα τοπικά ΜΜΕ και για το Radio Liberty. Ε, για το ότι ε, προσπαθούσε σκεφτεί πιθανούς λόγους για μια τρομοκρατική επίθεση στα γραφεία της FSB στην Βόρεια Ρωσία αντιμετωπίζει φυλάκιση 7 ετών. Ε, και αυτήν την έχουν αναλάβει οι δικηγόροι μας. Ε, θα τα δούμε αυτά στη συζήτηση. Αυτή η περίπτωση χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Όχι μόνο από τους Ρώσους υπεραστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά από ολόκληρη την ε, κοινωνία των πολιτών. Τελευταίο παράδειγμα. Ε, ΑΤΑΚ πριν από 10 μέρες ε, στην Τσετσενία. Πρόκειτο... για επίθεση στην Νόβα για Γκαζέτα, σε μια δημοσιογράφο της Νόβα για Γκαζέτα, την κυρία Μιλόσινα, η οποία κάλυπτε τα γεγονότα εκεί και τους επιτέθηκαν κάποιοι άνθρωποι στον Κρόσνη και μετά η κυρία Μιλάσενα η οποία δέχτηκε απειλές ε, στο email της μάλιστα στην εφημερίδα. Στην περίπτωση αυτή θα ζητήσουμε από την κυβέρνηση να ερευνήσει ουσιαστικά αυτές τις περιπτώσεις αλλά γνωρίζοντας το κλίμα ατιμορρησίας ε, και το της κοινή πρακτικής του ότι δεν ε, ερευνώνται οι επιθέσεις ούτε κάνει οι δολοφονίες δημοσιογράφων ε, φοβόμαστε ότι ούτε τώρα θα γίνει τίποτα. Αυτά. Θα μείνω σε αυτά τα ολίγα και έχω και κάποιες συστάσεις εάν θέλετε. Ευχαριστώ. Θα δώσω τον λόγο στον κύριο Τσαρνέτσκι κεφαλής αντιπροσωπείας ε, για την Ρωσία. Ε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, είμαι επικεφαλής αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τη Ρωσία και χαίρομαι για αυτή την ακρόαση. Όταν συγκριθεί με άλλες χώρες βλέπουμε ότι η Ρωσία δεν παίζει με τους κανόνες του παιχνιδιού. Δυστυχώς η συνταγματική αναθεώρηση δεν οδηγεί προς τη σωστή κατεύθυνση. Το Κρεμλίνο ε, θέλει να προωθήσει νόμους όπου μερικοί πολίτες ε, τίθενται υπεράνω άλλων. Επίσης, τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, τηρούνται μόνο στο μέτρο που επιθυμεί η κεντρική κυβέρνηση. Οι εκλογές δεν χάνονται ποτέ από τις δυνάμεις που υποστηρίζουν, στο, που υποστηρίζουν το Κρεμλίνο. Η Δούμα θέλει να αποδυναμώσει την κοινωνία των πολιτών και υπάρχει μεγάλη χρήση βίας και προωθούνται και οι νόμοι περί ξένων πρακτόρων, όπως είπατε και εσείς, το οποίο ε, αφορά οργανώσεις και φυσικά πρόσωπα. Η κατάσταση δεν θα βελτιωθεί υπό τον Πούτιν γιατί ε, ο εγχώριος νόμος είναι υπεράνω των, ε, του διεθνούς ε, δικαίου. Η προσάρτηση της Κρυμαίας επίσης μας απασχολεί ιδιαίτερα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε όλες αυτές τις ανησυχίες ήδη από πέρσι παρά την έλλειψη συναντήσεων με Ρώσους ομολόγους. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις στη Ρωσία πιστεύοντας ότι το συντομότερο δυνατόν θα ε, επαναπροσδιοριστεί ένας επικοδομητικός ε, διάλογος μεταξύ των δύο κοινοβουλίων. Η Ιζαμπέλ έχει το λόγο για το ΕΛΚ. Δίνω το λόγο στα μέλη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο ομιλητές μας ε, για τις εισηγήσει τους που ήταν πολύ λεπτομεριακές ε, και για να έχουμε μία καλύτερη εικόνα της κατάστασης μετά από όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Θα υποβάλω μερικές ε, ερωτήσεις. πώς ε, υπεραστίζεστε την ε, ελευθερία του, εκφράζεστε την ελευθερία του λόγου, γιατί η Ρωσία προβάλλει και διαδίδει ψευδείς ειδήσει. Πώς ε, τις αντιμετωπίζετε και πώς, ποια είναι η αντιμετώπιση στη Ρωσία. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Υπάρχουν πολλά μέλη, πολλοί ευρωβουλευτές που ανησυχούν διακόπτει η ομιλήτρια, έχει δυσκολίες μεταξύ Αγγλικών και Γαλλικών, όπως λέει η ίδια. Ωραία, βρήκα τη λέξη που ήθελα. Μιλάμε για απόπειρες να γραφτεί εκ νέου η ιστορία. Κάτι το οποίο θέτει πολλά προβλήματα. Πώς το βλέπετε εσείς ε, κατά τον ίδιο τρόπο που το βλέπουμε εμείς και πώς αντιδρούν οι πολίτες. Τέλος, ένα τελευταίο ερώτημα. Ποια είναι η άποψή σας για τις σχέσεις ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία. Πώς θα έπρεπε να προσδιοριστούν. Η Ευρώπη δεν είναι πάντα ενωμένη σε αυτό τον τομέα. Έχουμε αποκλίνουσες απόψεις από κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω όμως ότι θα έπρεπε να φτάσει σε μια κοινή θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς πώς βλέπετε το όλο θέμα. Ευχαριστώ. Ιζαμπέλ Σάντος για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Από τις δύο αυτές παρεμβάσεις, ε, από αυτές τις δύο μαρτυρίες, ανακύπτουν ορισμένα γεγονότα και συμπεράσματα. Υπάρχει έλεγχος της κοινωνίας, των ε, μέσων μαζικής ε, επικοινωνίας, των δημοσιογράφων και περιστέλλεται το δικαίωμα έκφρασης. Ένα λεπτό υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα με τη διερμηνία, γιατί δεν λειτουργούν σωστά τα συστήματα. Ωραία, θα ξαναρχίσω. Από τις δύο αυτές ε, μαρτυρίες για τη Ρωσία βλέπω ότι γίνεται μία απόπειρα ελέγχου της ρωσικής κοινωνίας, των ε, μέσων μαζικής ενημέρωσης, της κοινή γνώμης των ακτιβιστών και των δημοσιογράφων που αποτελούν μέσο διαμόρφωσης ε, της κοινή γνώμης. Όταν, ε, όταν ε, κυρώθηκε αυτός ο νόμος για τους ξένους, για τους ξένους ανταποκριτές, και τους ξένους πράκτορες θυμήθηκα την πρώην Σοβιετική Ένωση. Αυτό ήταν ε, ε, η σφραγίδα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Οι ΜΚΟ προσπάθησαν να δράσουν όσο μπορούσαν αλλά βλέπουμε ότι τώρα υπάρχει μία σοβαρή τροχοπέδη στη δράση τους καθώς και στη δράση των δημοσιογράφων. Αυτό μας απασχολεί γενικότερα και αφορά όλα τα απολυταρχικά καθεστώτα, ο έλεγχος της κοινή γνώμη και της ε, ελευθερίας λόγου. Και γι' αυτό ο κύριος Γιούση Λασίλα από ό,τι κατάλαβα και αν κατάλαβα καλά είπε ότι αυτή είναι μία αντίδραση της εξουσίας σε μία φάση που νιώθει ότι δεν εισακούεται Θεωρεί δηλαδή ότι χάνει τον έλεγχο η κεντρική εξουσία. Θα ήθελα να τον ακούσω και να μας μιλήσει και για την εξέλιξη της κοινή γνώμης και της ρωσικής κοινωνίας έναντι της εξουσίας. Ως προς την κυρία Αραπόβα, αναφέρθηκε σε δημοσιογράφους, σε ε, ακτιβιστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υφίστανται αντίπεινα και μην ξεχνάμε τον Αλεξέη Ναβάλνη που ήταν στο στόχαστρο του Πούτιν, ο κύριος στόχος του Πούτιν και θεωρήθηκε επίσης ξένος πράκτορας και φυσικά υπέστη αντίπεινα μέσα στα πλαίσια της τρομοκρατίας και του τρόμου αυτού. Αυτό είναι ένα μέσο δίωξης των δημοσιογράφων πολλές φορές. Θα ήθελα τις δικές σας υποδείξεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μας βοηθήσετε και να βοηθήσουμε αυτούς τους δημοσιογράφους που ζουν πολύ, πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα από αυτές τις διώξεις. Ευχαριστούμε. Ιζαμπέλ. Έχετε το λόγο από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, καθότι έχουμε τους ε, Κινέζους συνομιλητές μας στην οθόνη ακόμα, λέει η ομιλήτρια. Ε, βλέπουμε, ε, από ό,τι φαίνεται, ότι έτσι οι λάτρεις της απολυταρχίας αντιγράφουν ο ένας τον άλλον, λέει η ομιλήτρια χρησιμοποιούν δηλαδή κοινέ συνταγέ. Ευχαριστούμε την κυρία Ράποβα που μας τα εξήγησε όλα αυτά. Εγώ έχω μία-δύο ερωτήσεις. Νομίζω πέρυσι στις τοπικές εκλογές, αν δεν κάνω λάθος, το Σεπτέμβριο, είδαμε κάποια ενθαρρυντικά σημάδια τοπικών δημοκρατικών δυνάμεων που συνδέονταν με τοπικά κινήματα προστασίας του περιβάλλοντος νομίζω ότι είναι μια πολύ γνωστή περίπτωση, όχι εδώ, αλλά εκεί, σχετικά με την μεταφορά αποβλήτων από τη Μόσχα στο Αρχαγγέλσκ, στον Αρχάγγελο. Οπότε ήθελα να ρωτήσω και τον κύριο Λάσιλα και την κυρία Ράποβα μήπως υπάρχει μια νέα γενιά κοινωνικών κινημάτων που αμφισβητούν την εξουσία έτσι με εναλλακτικό τρόπο ίσως πιο επιτυχημένα. Η δεύτερη ερώτηση προς τον κύριο Λάσιλα, όπως είπε και η συνάδελφος για την, ε, το, το, το γράψιμο της ιστορίας εκ νέου και την ένωση για τη μνήμη ε, που έχει φυλακιστεί είδαμε ότι ε, πρόκειται να δοθεί αναστολή από το δικαστήριο μέχρι τις 10 ε, Φεβρουαρίου, δηλαδή πριν από λίγες μέρες. Πώς συνδέεται αυτή η περίπτωση σαν Ταρνόχα, αν ακούσαμε καλά, με αυτήν την, το νέο αφήγημα για την ιστορία. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική η περίπτωση και ελπίζω και οι ευρωπαϊκές αρχές να παρακολουθούν γιατί είχαμε μία δημοσιογράφος που είχε αναφέρει και επί του θανάτου κάποιων στρατιωτικών ε, πριν από κάποια χρόνια και τώρα μάλλον υποφέρει για αυτόν τον λόγο, για αυτά που είχε δηλαδή αναφέρει αποκαλύψει. Ευχαριστώ. Θα δώσω απευθείας το λόγο στον Γιούση πρώτα και μετά ε, και σε εσάς κυρία μου. Ευχαριστώ λέει ο κύριος Λάσιλα. Νομίζω ότι τα ερωτήματα ήταν συνδεδεμένα και θα έδινα μια αθρηστική απάντηση πρώτα. Ε, αναφερόμενος και στην λεπτομερή περιγραφή της κυρίας Σαράποβα και την όλο και μεγαλύτερη νομοθετική δραστηριότητα της κυβέρνησης προς πιο κατασταλτικά μέτρα. Νομίζω το θετικό σημάδι, μήνυμα, είναι αυτή η ατμόσφαιρα στην κοινωνία, στην κοινή γνώμη που αλλάζει και που συνδέεται και με το γεγονός ότι όλη αυτή η κατασταλτική νομοθεσία και τα μέτρα δεν είναι μια ιδεολογική προσέγγιση από το καθεστώς λέει ο μιλητής αλλά αντίδραση έναντι της, ε, του εύθραυστου της εξουσίας τους όπως το αντιλαμβάνονται. οι προηγούμενες αντιδυτικές ή συντηρητικές ή δεν ξέρω πώς να τις αποκαλύψω μη φιλελεύθερες προσεγγίσεις δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές για την κοινή γνώμη και η μεγαλύτερη δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένια, Ευρω... Ε, Ένωσης με είναι ότι αυτές οι φιλελεύθερες αξίες λέει ο μιλητής χαίρουν ακόμα μεγαλύτερης αναγνώρισης στη Ρωσία σήμερα. Γιατί από ό,τι φαίνεται οι πολίτες αντιστέκονται σε αυτές τις ιδέες που θέλει να τους επιβάλλει το καθεστώς. Αν ξαναδούμε την ατμόσφαιρα που επικρατούσε από το 14 στο 16, όπου υπήρχε μια πολύ σημαντική συνένεση και έτσι πατριωτική εφορία, το κατόφλι της εισαγωγής τέτοιων νομοθετικών διατάξεων θα ήταν πολύ υψηλότερο. Βέβαια είναι τόσο αδύναμη η οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών και η εκπροσώπηση της που το καθεστώς έχει ευκαιρίες να υλοποιήσει, αλλά πρέπει να λαμβάνει υπόψη του πιθανές αντιδράσεις. Και αυτά που είπε και η κυρία Χάουταλα, αυτές οι αναφορές στα οικολογικά θέματα, αυτό είναι μια νέα διάσταση στην στο ρωσικό δημόσιο βίο. Ίσως όλα αυτά δείχνουν απλώς ότι η Ρωσία αφυπνίζεται περιβαλλοντικός μιλώντας. Ακόμα και συζητήσεις για την κλιματική αλλαγή γίνονται, λέει ο μιλητής. Και είχαμε και διαδηλώσεις κατά ε, συγκεκριμένων τόπων που χρησιμοποιούνταν ως χωματερές. Ε, Στο Εκάτεριμπουργκ υπήρχε τοπική διαδήλωση κατά του Ορθόδοξου Ναού που επρόκειτο να οικοδομηθεί στην κεντρική πλατεία. Ε, η αντίδραση ήταν τέτοια που το σχέδιο ανεβλήθη όπως και η περίπτωση Γκολούνοφ. Τώρα, πώς αντιδρούν στη Ρωσία σχετικά με τα λεγόμενα fake news νομίζω το επίπεδο ψευδούς ενημέρωσης μάλλον λίγο υπερβολικά αποτυπώνεται στα δυτικά μέσα λέει ο μιλτής η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ μεγαλύτερη ήπια δύναμη soft power για να το πούμε ελληνικά από ότι η Ρωσία. Ε, αναγκάζονται να χρησιμοποιούν κατασταλτικά μέσα γιατί δεν έχουν και πολλά άλλη μέσα στη διάθεσή τους γιατί ε, δυσκολεύονται να βρουν, να εξεύρουν ένα πιο φιλελεύθερο μέσο ή λύση. και δυσκολεύονται να περιγράψουν, αν θέλετε, μια ευνοϊκή στάση της κοινωνίας απέναντι σε αυτήν την απόπειρα της επανασύνταξης της ιστορίας. Δηλαδή βλέπουμε κάποιες αλλαγμένες, ε, τροποποιημένες τάσεις για τον τρόπο που αναφερόμαστε παλαιότερα ιστορικά περιστατικά, όπως και την καταστολή υπό το Στάλιν, που τώρα συνοδεύεται και από τα θετικά της χαρακτηριστικά. Um, ναι, ναι. Μάλιστα. Ευχαριστώ για τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Πολύ σημαντικές όλες. Δεν ξέρω αν μπορώ να τις απαντήσω όλες, αλλά θα προσπαθήσω. Εγώ είμαι δικηγόρος, ε, υπερασιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν είμαι πολιτικός. Οπότε κάποιες απόψεις που θα εκφράσω θα είναι είτε προσωπικές ή αυτή με την οποία συμφωνούν και οι συναδελφοί μου. Πρώτα απ' όλα, διάδοση ψευδών ειδήσεων και το αν ε, η προπαγάνδα είναι αποτελεσματική. Εγώ θα συμφωνήσω με τον καθηγητή Λασίλδα ότι δεν είναι τόσο αποτελεσματική πια. Η νέα γενιά ε, που ενημερώνεται στο διαδίκτυο ε, δεν επηρεάζεται από την προπαγάνδα αυτή των τηλεοπτικών σταθμών. Υπάρχουν βεβαίω ε, τα τρόλ του Κρεμλίνου, αλλά δεν είναι τόσο προχωρημένα και η νέα γενιά δεν θεωρεί ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να εμπιστευτεί. Οπότε έχουμε τώρα την αύξηση της νέας γενιάς που διαμαρτύρεται για το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, για το δικαίωμα διάδοση πληροφοριών. Και βεβαίως ε, είναι εύκολο να δούμε ποιες είναι οι πηγές της προπαγάνδας ε, και να τις κατονομάσουμε, να τις στιγματίσουμε αν θέλετε. Είναι θέμα ενημέρωσης δηλαδή περί των θεμάτων των ΜΜΕ για να ξέρει ο κόσμος ποιες πηγές μπορεί να εμπιστεύεται, ποιο είναι πίσω από μια πηγή πληροφόρηση. Γιατί εμφανίζονται διάφορα κανάλια στην εφαρμογή Telegram, ε, πολύ σημαντικά για όσους πληροφορούνται από το διαδίκτυο και δεν είναι πάντα σαφές ε, ποιος τα ελέγχει. Μια φορά τα ελέγχουν αυτές οι αρχές, αλλά προσπαθούν να το παίξουν ε, φιλελεύθερα. Οπότε... Το θέμα είναι πώς θα είναι αυτά προσβάσιμα στη Ρωσία χωρίς να μπλοκάρονται. Η Ρωσία θα έχει πρόσβαση σε αυτές τις ε, πληροφορίες. Λοιπόν, όσον αφορά ε, την ιστορία και την ε, συγγραφή της, δεν ξέρω πώς να το προσεγγίσω γιατί δεν βλέπω ότι η ρώσικη κοινωνία έχει κάποια απάντηση σε αυτά τα ζητήματα. Δεν είναι ένα θέμα που απασχολεί τα ρωσικά μημιέ. Τα ανεξάρτητα μίμιε το θίγουν, ε, λένε ότι είναι ένα είδος ε, προπαγάνδας ε, το οποίο δεν είναι πάντα κατάλληλη, αλλά νομίζω ότι το ζήτημα αυτό ενδιαφέρει τη νέα γενιά. λένε τους χάρη ναι, ναι, ποιος ξεκίνησε το δεύτερο παγκόσμιο και τα σχετικά. Λοιπόν, η δημόσια συζήτηση και η ελεύθερη ροή πληροφοριών είναι πάρα πολύ σημαντική. Και βέβαια και η εμπειρογνωμοσύνη από διάφορα μέρη του κόσμου έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Το τελευταίο ζήτημα οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι η περίπτωση του κυρίου Δημητρίευ και η επίθεση στα γραφεία της οργάνωσης Memorial ε, είναι στις γενικότερες επίθεσεις επίθεσης της ΜΚΟ Είναι λοιπόν ε, η Memorial μια οργάνωση κλειδί η οποία πάντα είναι στο στόχαστρο. Τώρα έχουν στόχαστρο 6 εκατομμυρίων ρουβλίων γιατί δεν ανεβάζουν όλες τις θέσεις στο διαδίκτυο. Ε, είναι στο πλαίσιο της ευρύτερης εκστρατείας θα έλεγα. και εδώ πρέπει να βοηθήσουν όλοι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομίζω.